Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς Θα το γυρίσω στη μητρική μου γλώσσα που είναι τα Ουγγρικά. Ε, Καλημέρα σας λοιπόν και Ουγγριστή. Καλωσορίζουμε τα μέλη της Επιτροπής μας στην Επιτροπή Αναφορών. Καλωσορίζουμε τα μέλη μας, τους αναφερομένους, τους εκπροσώπους τους, όλους εκείνους που εκπροσωπούν την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γενικότερα τους προσκεκλημένους μας και τους επισκέπτες. Σας ζητώ συγγνώμη, διότι είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που προεδρεύω. σε συνεδρίαση Επιτροπής. Οπότε μπορεί να έχω κάποιες αβεβαιότητες και ανασφάλειες ως προς τα διοικητικά και τα θέματα της γραμματείας και προσβλέπω στη γραμματεία για να με βοηθήσει στην προσπάθεια αυτή. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα ως πρώτο θέμα έχουμε σημαντικό έγγραφο εργασίας της κυρίας Γούλης. Ελπίζω να το γνωρίζετε. Και θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Γόλης, που είναι η συγγήτρια, να λάβει το λόγο και να μας κάνει την εισαγωγή της. Παρακαλώ, κυρία Γόλης. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Συγχαρητήρια για την παρθενική σας Προεδρία. Το πρόγραμμα της Στοχόλμης. Αν μου επιτρέψετε, θα ήθελα να χωρίσω σε τρία τμήματα την ε, παρουσίασή μου. Πρώτα, τι κάνει το Κοινοβούλιο, στη συνέχεια ε, την ουσία του θέματος και το τρίτο είναι το έγγραφο εργασίας. Πρώτο, η διαδικασία. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να γνωμοδοτήσει για το πρόγραμμα της Στοχόλμης, που είναι και πρόγραμμα της ε, Προεδρίας αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έλεγα πρέπει να γνωμοδοτήσει το Κοινοβούλιο σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα. Τρεις είναι οι βασικές επιτροπές καθήλυνα αρμόδιες που προετοιμάζουν έκθεση ε, και ψήφισμα και είναι η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, Πολιτικών Ελευθεριών και η Νομική η δική μας Επιτροπή συμμετέχει μεν, αλλά ως γνωμοδότηση μόνο είτε η δική μας συμμετοχή και θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα συμπεριληφθεί ε, στο σύνολο των άλλων εκθέσεων και δική μας ε, γνωμοδότηση. Στη συνέχεια θα έρθω στα γράμματα. Εμείς έχουμε λοιπόν σε αυτό το στάδιο ένα έγγραφο εργασίας, το οποίο έχουν λάβει και έχουν στα χέρια τους αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας πω το εξής για το πλαίσιο. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είναι ένα πρόγραμμα πενταετές στον τομέα της ασφάλειας και της αστικής δικαιοσύνης. Και ακολουθεί άλλα πρόγραμμα. Το προηγούμενο μας ήταν πρόγραμμα της Χάγης και το προπροηγούμενο πρόγραμμα του Τάμπερε. Αυτό που έχει σημασία να πούμε τώρα για τα έγγραφα και τις προσδοκίες που έχουμε για την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι αν ε, τρέξουμε στο 1999 θα θυμηθούμε ότι υπήρχε σαφής βούληση από τότε να γίνουν κάποια βήματα στη δικαιοσύνη για να ε, βοηθήσουμε τους πολίτες στην καθημερινή του ζωή. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου όμως άλλαξαν τα πράγματα και δόθηκε πολύ περισσότερη έμφαση στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και στα θέματα ασφαλείας, όπως θα ήταν και αναμενόμενο άλλωστε. Τώρα όμως έχουμε ξανάρθει σε ένα σημείο ε, που υπάρχει ευκαιρία να ε, ε, εξισορροπήσουμε και πάλι τη σκέψη μας και να ε, στραφούμε πιο πολύ στους πολίτες και στην καθημερινότητά τους και στα δικαιώματά τους. Αν κοιτάξετε λοιπόν και το έγγραφο της Σουηδικής Προεδρίας αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ εστιασμένα τα κείμενα στα δικαιώματα των πολιτών, στην ενίσχυση, στην ενδυνάμωσή τους και στη διεκδίκησή τους μέσω των δικαστήριων. Όλη η προσέγγιση λοιπόν είναι υπέρ του πολίτη. Νομίζω υπάρχει και ένα σύνθημα να βάλουμε τον πολίτη στο κέντρο της Ευρώπης. Ξέρω ότι τα έχουμε ξαναπεί και ξανακούσει όλα αυτά ε, ξανά και στο παρελθόν, αλλά ακόμα και εγώ είμαι κάπως αισιόδοξη ότι πραγματικά βρισκόμαστε τώρα σε καλό δρόμο και θα κάνουμε πρόοδο. Βεβαίως τα δικαιώματα των πολιτών και η ενίσχυση των πολιτών για να μπορέσουν να τα διεκδικήσουν και να, τα, και να δικαιωθούν είναι πάγια υπόθεση και εργασία της Επιτροπής μας. Γι' αυτό θα πρότεινα να κοιτάξουμε τι κάνουμε τώρα στην Επιτροπή που έχουμε πολλές αναφορές που ασχολούνται και ε, αφορούν και αντικατοπτρίζουν το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, δηλαδή να προσθέσουμε κάποιο ειδικό βάρος και να τονίσουμε την ανάγκη ότι αυτά τα θέματα πρέπει να προωθηθούν και να δοθεί συνέχεια. Στο έγγραφο λοιπόν εργασίας έχω τονίσει συγκεκριμένους τομείς. Η πλήρης άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας. Ε, Έχουμε πάρα πολλέ αναφορές πολίτων. Η προστασία των ανηλίκων. Έχουμε ε, ε, και ειδικά θέματα που απασχόλησαν την Επιτροπή μας. Συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή τη Ένωση. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν. Και ελπίζω ε, επίση να βγει και κάτι από τη Λισαβόνα που μας ενδιαφέρει πολύ, που είναι η πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών. Και είναι σωστό να το λέμε και στο κείμενο εργασία ω Επιτροπή θέματα που έχουν να κάνουν με την αμοιβαία αναγνώριση από εκεί και πέρα και πολιτική θεώρηση διαβατήρια. Όλα αυτά τα θέματα ε, μας δείχνουν ότι υπάρχουν προβλήματα για τους πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε την εμπειρία από την Επιτροπή μας για να δούμε αυτά τα θέματα. Βεβαίως, πολλά από τα ζητήματα αυτά δεν χρειάζεται μια νομοθεσία. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Συχνά χρειάζεται καλύτερη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Και θα το βρείτε και αυτό και στα συμπεράσματα και στις συστάσεις μου. Τονίζουμε ότι χρειάζεται καλύτερη ε, εφαρμογή και εκεί είναι το μέγα πρόβλημα. Και το πρόγραμμα της Οχόρμης θα πρέπει να ασχολείται με αυτό. αν θέλουμε πραγματικά να, έχουμε, να παρέχουμε στους πολίτες μας τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια που επιθυμούν. Αυτά. Σύντομα ως προς τον προσανατολισμό του κειμένου, όπως προσπάθησα να σας πω στην αρχή, έχουμε κάποια χρονική πίεση για να βεβαιωθούμε ότι θα ακουστεί και η δική μας φωνή ως Επιτροπής Αναφορών. Οι τρεις καθήλυνα αρμόδιες επιτροπές ήταν επιτροπές που θα κάνουν ε, την έκθεση του 8 Οκτωβρίου και η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι 22 Οκτωβρίου. Αλλά αν θέλουν οι πολίτες να δεχτούμε αυτό το κείμενο, νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια τέτοια διαδικασία και θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ακριβώς οι απόψεις μας θα συμπεριληφθούν στο κείμενο. Τελικά λοιπόν μπορούμε να πούμε και πρέπει να πούμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη πρακτική εμπειρία η Επιτροπή μας για να βοηθήσει στη διαμόρφωση του προγράμματος της Στοκχόλμης. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να σας βοήθησε το έγγραφο εργασίας μου προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος, για τις παρατηρήσεις σας αυτές για ε, τις επιτροπές και τις εργασίες μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το έγγραφο αυτό ασχολείται με τις αντιφάσεις που υπάρχουν, δηλαδή και είναι μεγάλη πρόκληση για τον 21ο αιώνα. Από τη μια η ασφάλεια, το οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία, αλλά και η προστασία των πολιτών, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Εκεί θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Γι' αυτό συμμετέχουν πολλές ε, επιτροπές σε αυτό το εγχείρημα. Η Επιτροπή Ελευθεριών ασχολείται κατά κύριο λόγο, αλλά είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα. Και τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν θέλει να πάρει το λόγο. Ναι, ναι, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ και εγώ για την παρθενική σας εμφάνιση στην Προεδρία της Επιτροπής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα την κυρία Γόλης για την έκθεσή της. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και περιγράφει τέλεια και απόλυτα τις προθέσεις της Ευρω... και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα της Στοχόλμης. Θα ήθελα να σας δώσω μερικά ε, γενικά στοιχεία πριν μπω σε λεπτομέρειες. Πρώτον, για το πρόγραμμα έγκρισης η Σουηδική Προεδρία έχει μπει τώρα σε σημαντική φάση διαπραγματεύσεων, διαβουλεύσεων για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να εγκριθούν ε, οι συστάσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 10ης Δεκεμβρίου. Μετά το πρόγραμμα της Στοχόλμης θα ακολουθήσει ένα πρόγραμμα δράσης που συγκεκριμένα θα περιγράψει όλες αυτές τις δράσεις ε, που θα πρέπει να υλοποιηθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει σίγουρα προτάσεις τέλη του ε, χειμώνα για να εγκριθεί τον Ιούνιο στο Συμβούλιο στην Ισπανική Προεδρία. Ε, η διαδικασία αυτή θα κρατήσει κάποιο διάστημα υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί στόχοι που θα πρέπει να ε, τεθούν και από εκεί και πέρα συγκεκριμένες δράσεις στα θεσμικά όργανα και στα κράτη-μέλη. Τώρα, επί της ουσίας, θα πρέπει να σας πω ότι διαβάζοντας την έκθεση της κυρίας Γόλης, αισθανθήκα μεγάλη ικανοποίηση, διότι ακριβώς ε, καταδεικνύει αυτό που θέλουμε εμείς και αυτό που θέλουμε να βελτιώσουμε στο πρόγραμμα αυτό στο Χόλμες. Το εξήγησε επανειλημμένα αυτό ο Αντιπρόεδρος Μπαρό, κατά τα άλλα. Τώρα που τα θέματα ασφάλειας, δικαιοσύνης και ελευθερίας ε, είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας τα τελευταία δέκα χρόνια, θα πρέπει να τα ξαναδούμε γιατί ε, φύγουν ε, την καθημερινή ζωή των πολιτών και μάλιστα τους αφορούν πάρα πολύ άμεσα. Ε, πολύ ωραία τα περιγράφει η εκθέση της κυρίας Καθημερινά οι πολίτες αντιμετωπίζουν μια σειρά ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τις πολιτικές αυτές. Σήμερα υπάρχουν ορισμένες τάσεις οι οποίες έχουν αρχίσει να χαράζονται στα πλαίσια του μελλοντικού προγράμματος της Στοχόλμης και η έκθεση προς την κατεύθυνση αυτή κινείται. Καταρχήν δίδεται μεγάλη σημασία στην εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων. Έχει υπάρξει αρκετά σημαντική νομοθετική δουλειά τα τελευταία δέκα χρόνια. Έχει υπάρξει ένα ουσιαστικό και εκτιμένο, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί σίγουρα σε ορισμένους τομείς. Αυτό όμως το οποίο χρειάζεται είναι η εφαρμογή θα πρέπει να συνοδευτεί η εφαρμογή αυτών των μέσων. Ξεκίνησε να το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της οδηγίας 2004-38 για την ελευθερία διακίνησης. Έχει δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχουν σαν στόχο τη διευκόλυνση της εφαρμογής της οδηγίας αυτής. Μια οδηγία η οποία μας απασχολεί ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί οι μισές διαδικασίες επί παραβάση αφορούν τη συγκεκριμένη οδηγία. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να γίνει στον τομέα της βελτίωσης της εφαρμογής της οδηγίας και μια ολόκληρης σειρά παράλληλων επίσης μέτρων. Είδαμε χαρά ότι υπογραμμίζεται το θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης των ληξιαρχικών πράξεων είναι σαφές ότι μας περιμένει πρόοδος τα επόμενα χρόνια. Είναι δύσκολος ο τομέας γιατί υπάρχουν εντελώς διαφορετικές ευαισθησίες στο συγκεκριμένο. Δεν θα πρέπει να είναι δύσκολο όταν έχουμε μια ληξιαρχική πράξη από μια χώρα να γίνει αντικείμενο αναγνώρισης από μια άλλη. Ένα άλλο θέμα το οποίο συμπληρώνει τις παρατηρήσεις μου. Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να διαφθρώνονται και με άλλες μορφές πολιτικής. Το βλέπουμε σαν παράδειγμα σε αυτά τα οποία λέγονται για την προστασία των ανηλίκων. Η προστασία την οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προβλέπει ένα νέο πλαίσιο για την προστασία των ανηλίκων και διασταυρώνεται αν θέλετε και με κάποια μέτρα της δικής μας πολιτικής βελτιώνοντας τα μέντα δε. Μια παρατήρηση γενικού ενδιαφέροντος. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διατυπώθηκε για να είναι όπως ονομάζουμε Lisbon Neutral, δηλαδή να μην εξαρτάται από την τύχη της συνθήκης. Προβλέπουμε ορισμένους στόχους οι οποίοι ε, μπορούν να στοχευθούν ακριβώς ε, και ανεξάρτητα από την τύχη της συνθήκης της Λισαβόνας. Θα γνωρίζουμε περισσότερα σε λίγες μέρες βέβαια. Πάντως μια ολόκληρη σειρά πολιτικών δράσεων θα πρέπει να διευκολυνθεί. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριο Γόλες για την έκθεσή σας, να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο γενικότερα, την Σουηδική Προεδρία η οποία εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά για την διαμόρφωση του προγράμματος της Στοκχόλμης. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω τώρα από την συντονίστρια αν θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, λέει η κυρία Γκρινή. Ευχαριστώ και την κυρία Γόλης για αυτό το κείμενο εγγρασίας. Δεν το έχουμε στις γλώσσες μας μεταφρασμένο και αυτό είναι λίγο δύσκολο. Πάντως θα πρέπει ο πολίτης να βρεθεί στο κέντρο των ανησυχιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι η ουσία. Και βλέπουμε μάλιστα στα πλαίσια της Επιτροπής Αναφορών και των αναφορών που φτάνουν ότι το συγκεκριμένο θέμα παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον. Το θέμα της αναγνώρισης του γάμου ανάμεσα σε πρόσωπα ιδίου φύλου. Αυτό είναι κάτι το οποίο ανήκει πάντα στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Είναι δύσκολο θέμα. Εγώ ήμουν μέλος της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και έχουμε συζητήσει πολύ το πρόβλημα γιατί πίσω ακριβώς από τον γάμο των ομοφιλοφίλων υπάρχει μια ολόκληρη προβληματική για την ε, ομογονεϊκότητα και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και μας απασχολεί. Στη Γαλλία λύσαμε το πρόβλημα μέσω του λεγόμενου συμφώνου, γαμικού συμφώνου του ΠΑΞ και λύσαμε και τα προβλήματα τα κληρονομικά και διαδοχής και τα λοιπά, αλλά υπάρχουν άλλα χαίνοντα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτές οι συνεισφορές ε, αναφέρθηκαν στα δικαιώματα στην ελευθερία και για την ασφάλεια. Όλα αυτά ήταν νέα στοιχεία και κοιτώ προς την πλευρά του κυρίου. David, από εσά εξαρτάται πλέον, από τα μέλη του Κοινοβουλίου, από τα μέλη της Επιτροπής αυτής, να θέσουν ερωτήματα, να κάνουν τις σωστές ε, συνεισφορές, τις σωστές συμβολές. Σε αυτή τη φάση νομίζω λοιπόν ότι έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν σχόλια, θα ήθελα να δώσω το λόγο και πάλι στην εισηγήτρια, στην κυρία Βόλης. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Φαίνεται ότι η Επιτροπή στηρίζει την προσέγγισή μας και χαίρομαι για τα σχόλια που άκουσα. Αν αυτό είναι το γενικό πλαίσιο και η γενική αίσθηση που επικρατεί, ελπίζω να μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Λυπάμαι που δεν υπάρχουν μεταφράσει ακόμα, αλλά ήταν και στενά το χρονοδιάγραμμα. Μπορεί να ακολουθήσουμε όμως από ό,τι κατάλαβα μια γραπτή διαδικασία και η γραμματεία θα μπορούσε ίσως να μας εξηγήσει ποια θα είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει στην περίπτωση αυτή. Η γραμματεία είναι σε επαφή με τις ε, βασικές, ε, με τις τρεις αρμόδιες επιτροπές προκειμένου να συντονίσουμε την ε, συνεισφορά μας ως Επιτροπή. Αλλά προφανώς όλα εξαρτώνται από το σχέδιο ψηφίσματος. Αυτό ακόμη δεν διατίθεται. όταν θα το έχουμε στα χέρια μας θα το μοιράσουμε σε όλα τα μέλη της Επιτροπής και θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι στις 19 Οκτωβρίου θα γίνει έκτακτη συνάντηση της Επιτροπής μας στο Στρασβούργο όπου μπορεί να έχουμε άλλα προβλήματα αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να κοιτάξουμε και πάλι το θέμα αυτό. Ωστόσο, όταν θα έχουμε τα σχέδια ψηφισμάτων από τις άλλες επιτροπές θα τα διαβιβάσουμε στα μέλη και βάσει των σχεδίων αυτών θα έρθουμε σε επαφή με τις διάφορες ε, ομάδες και μετά θα καταρτιστούν ε, ενδεχόμενες φροπολογίες. Ελπίζω να μην είναι πολλά στον αριθμό, οι οποίες θα εγκριθούν από τους συντονιστές των ομάδων. Και έτσι λοιπόν ε, αυτή τη διαδικασία θα ακολουθήσουμε ιδάλλως στις 3 και 4 Νοεμβρίου που θα είναι η μεθεπόμενη συνάντηση της ομάδας θα είναι πολύ αργά Άρα θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπημένη λύση που θα επιτρέψει την συμβολή από όλες τις ομάδες και να αποφασίσει τελικά με ποιο τρόπο θέλουμε να προχωρήσει η Επιτροπή. Έχουμε με την έγκριση της κυρίας Βόλησε ήδη διαβιβάσει το σχέδιο προς τις ε, ομάδες εργασίας και σε ό,τι αφορά τις ε, μεταφράσεις όταν θα τις έχουμε στη διάθεσή μας, θα τις στείλουμε κατευθείαν μέσω email στην Επιτροπή, προκειμένου να έχετε ο καθένας το έγγραφο στην γλώσσα του. Μάλιστα, λέει η Πρόεδρος. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Γουόλης και όλους όσοι έκαναν σχόλια για τις παρατηρήσεις τους. Ολοκληρώνεται λοιπόν η συζήτηση του θέματος αυτού και ελπίζω να έχουμε χρόνο όλοι να διαβάσουμε το έγγραφο, να ασχοληθούμε με αυτό και θα συνεχίσουν ε, θα, συνεχίσει, συνεχιστεί η εξέταση σε όλες τις πολιτικές ομάδες προκειμένου κάθε ομάδα να καταλήξει στις ανάλογες συστάσεις. Και τώρα να συνεχίσουμε με τις αναφορές σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική προστασία καταρχάς. Να συζητήσουμε καταρχάς την ε, αναφορά 650-2008 του κυρίου Μπίλι Λέοναρτ από την Ιρλανδία. Είναι εδώ? Καλώς ήρθατε λοιπόν. Να δώσω λοιπόν το λόγο κατευθείαν στον κύριο Λέοναρντ. Πέντε λεπτά. Please, Mr. Ε, thank you. Ο κύριος Νέλναρντ, ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας ε, συγχαρώ για τη νέα σας θέση. Είμαι τοπικό σύμβουλος στο Κολορίον και αυτό σχετίζεται με την ε, αναφορά αυτή. Πρόκειται για μια πολύ μικρή κοινότητα, η οποία είναι αντιμέτωπη με μια τεράστια εγκατάσταση. Σας έχω δώσει κάποιες ε, πληροφορίες για το ιστορικό και έχουμε δώσει και επιχειρήματα για, το, για τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που δεν τηρούνται και όταν έγραψα στον κύριο Λόου την 1η Απριλίου του 2009. Νομίζω ότι τα έχετε αυτά τα στοιχεία, δεν θα ήθελα να τα επαναλάβω λοιπόν και να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Μιλάμε λοιπόν για εγκαταστάσεις ε, επεξεργασίας απορριμμάτων σε μια πολύ μικρή κοινότητα. Δεν ε, πρόκειται, θα ήθελα να διευκρινίσω, για κάτι το οποίο δεν θέλουμε απλά να εγκατασταθεί στην ε, δική μας περιοχή. Μιλάμε για μια περιφέρεια που έχει χιτά εδώ και καιρό και ε, αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα από τον τρόπο λειτουργίας των χιτά αυτών. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να τονίσω ότι δεν πρόκειται για μια περίπτωση όπου μια κοινότητα δεν θέλει να λάβει τις ευθύνες της και απλά θέλει να διώξει μια τέτοια εγκατάσταση. Όχι. Υπάρχει μια ενεργή εγκατάσταση στην περιοχή, στο Greg Road, και σημειώθηκαν πολλά περιστατικά κακής πρακτικής ε, στο, στην περιοχή αυτή και έγιναν και έρευνες ε, του λαβετή. Έκλεισαν ε, κάποιες εγκαταστάσεις και ο, προ, ο πρώην ιδιοκτήτης μπήκε στη φυλακή. Γενικώ η ιστορία είναι αρκετά βεβαρημένη, το ιστορικό. Η όλη διαδικασία αυτή και η όλη δικαστική αγωγή έλαβε χώρα το 2006 και αποφασίστηκε τότε ότι δεν χρειάστηκε διαδικασία, πλήρη διαδικασία για υποβολή αίτηση. Για την κατασκευή δηλαδή, τα οικοδομικά έργα. Τότε λοιπόν το 2006 αναφέρθηκε ότι ουσιαστικά δεν υπήρχε και ανάγκη να γίνει οποιαδήποτε περιβαλλοντική ε, μελέτη. Άρα, μιλάμε για μια μεγάλη έκταση που θα χωράει 200.000 τόνους ανά έτος και πρότυπα 30 κονταετίας ουσιαστικά του 1976 για μια τέτοια εγκατάσταση που επανεκκινεί τη λειτουργία της και η κοινότητα αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα, έχει πάρα πολύ άσχημη εντύπωση από το γεγονός ότι δεν έγινε σχετική μελέτη. Επίσης, προσφάτως έγινε αίτηση για αύξηση ε, του όγκου και των ειδών απορριμμάτων που υπόκεινται επεξεργασία. και πάλι δεν έγινε η σχετική πλήρης αίτηση. Ο υπουργό φαίνεται ότι άλλαξε γνώμη και τώρα ζητά να υποβληθεί επίσημη πλήρης έταση, ε, αίτηση. Άρα φαίνεται ότι η πίεση από τη κοινή γνώμη ε, απέφερε καρπούς. Μιλάμε για εγκαταστάσεις οι οποίες ε, θα επεξεργάζονται 500.000 τόνους το έτος και 600.000 τόνους το έτος. Αλλά μία από τις εγκαταστάσεις αυτές παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα και αυτό ε, σε όλα αυτά σε μια περιοχή ιδιαίτερη φυσικού κάλους επηρεάζει φυσικά την άγρια πανίδα και χλωρίδα και μιλάμε για πλούσια πανίδα, πολλές, ε, πολλά είδη για παράδειγμα λαγών, κουνελιών, πεταλούδων και λόγω του κακού ιστορικού επειδή υπάρχουν αυτές οι ελλειπεί αιτήσει, ζητούμε η Επιτροπή Αναφορών να ελέγξει ότι εφαρμόζονται τα πρότυπα της Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση αυτή. Και για παράδειγμα, έγραψα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντας και ζήτησα πριν από την ακρόαση αυτή να μας πει πώς το Υπουργείο ε, ανταποκρίνεται, πώς θεωρεί ότι αντιρούνται τα πρότυπα των ε, οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην απάντησή του δεν αναφέρεται σε καμία από τις οδηγίες αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια, τα κριτήρια, τα μέτρα που θέτουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες δεν εφαρμόζονται όπως θα έπρεπε κατά την εφαρμογή και την επεξεργασία των αιτήσεων αυτών που υποβάλλονται. Γι' αυτό λοιπόν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε την αίσθηση ότι ήταν μάλλον σε πρώτη φάση η υποβολή του αιτήματό μας. Όχι, θεωρούμε ότι επειδή βρίσκονται σε φάση επεξεργασίας αυτές οι αιτήσει, τώρα θα πρέπει να κοιτάξουμε τον αντίκτυπο. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Επιτροπή Αναφορών να συνεχίσει να εξετάζει το θέμα αυτό και το αίτημά μας. Και ξέρω ότι σίγουρα ο κόσμος στην περιοχή μας θα είναι πάρα πολύ ευγνώμων για την αντιμετώπιση αυτή. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Είναι σαφή ε, η επιχειρηματολογία σας και όλοι μας ανυπομονούμε να ακούσουμε την γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να στραφώ λοιπόν προς τον κύριο Πάτης. Δεν ξέρω αν βρίσκεται εδώ. Ε, thank you, ε, Mrs. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Είμαι ο κύριος Δίας, όχι ο κύριος Πάτης. Γιατί ουσιαστικά δύο νομοθετήματα εμπλέκονται εδώ. Η οδηγία για τις χωματηρές και η άλλη οδηγία για τη μελέτη αντικτύπου. Εγώ είμαι υπεύθυνο για την οδηγία για τους χώρους υγειονομικής ταφής και ο συνάδελφός μου θα αναφερθεί πιο πολύ στη, για την οδηγία για τη μελέτη αντικτύπου, περιβαλλοντικού αντικτύπου. Το παράρτημα 1 για την ε, οδηγία για τους χιτά του 91, 99, κάθετος 31, θέτει τις παραμέτρους για όλους τους χιτά, μεταξύ των οποίων και η τοποθεσία τους. Και αυτό εναπόκειται στις εθνικές ε, αρμόδιες αρχές, υπό τον όρο ότι δεν εμπλέκονται σημαντικοί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι. Στα πλαίσια της οδηγίας δεν τίθενται συγκεκριμένοι όροι για τις αποστάσεις που θα πρέπει να τηρούνται μεταξύ των διαφόρων χιτά. Και να αναφέρω και ένα πολύ σημαντικό άλλο άρθρο, το άρθρο 7 της οδηγίας για την υποβολή αιτήσεων για έγκριση, που θα πρέπει να περιέχει μελέτη αντικτύπου αν πρόκειται για χιτά που περιλαμβάνεται στο, στην οδηγία 85 κάθετος 337, όπως έχει τροποποιηθεί. όπου αναφέρεται ο κοινωτικό αντίκτυπο και όπω σα είπα, ο συναδελφό μου είναι πλέον αρμόδιο για τέτοια θέματα. Σύμφωνα με τι πληροφορίε που έχουμε λάβει ω τώρα, φαίνεται ότι είναι ακόμα πολύ νωρί για να θεωρήσουμε ότι υπάρχει παραβίαση της οδηγίας για τους χιτά. Άρα, ο αναφερόμενος θα έπρεπε να παρέχει επιπλέον πληροφορίες για να αποδείξει κακοδιαχείριση της ε, εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή θα χαρώ να κοιτάξω και να εξετάσω σε βάθος το διαχειριστικό αυτό σκέλος σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση της οδηγίας για τους χιτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει τα δέοντα μέτρα. Αυτά λοιπόν. Και όπως σας είπα, εγώ μιλάω για την οδηγία για τους χιτά. Ο συνάδελφος θα μιλήσει για την οδηγία για τη μελέτη αντικτύπου. Ευχαριστώ πολύ. Σε ό,τι αφορά την οδηγία για το, τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, την 85335, έχουμε δύο πτυχές. Καταρχάς, το σωρευτικός αντίκτυπος κάποιων εγκαταστάσεων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν αποφασίζουμε κατά πόσο χρειάζεται μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε για την εγκατάσταση του Camp Road, υπάρχει αίτηση πλήρης από το Μάρτιο του 2009 με μελέτη αντικτύπου. Άρα υποθέτουμε ότι ο σωρευτικός αντίκτυπος ε, θα ληφθεί υπόψη και θα εκτιμηθεί σε ό,τι αφορά τα άλλα δύο project, τα άλλα δύο έργα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε, δεν υπάρχει ακόμα τέτοια αίτηση. Υποθέτουμε ότι θα ληφθούν υπόψη όλες οι κατάλληλες παράμετροι και θεωρούμε ότι οι αρχές της Βορείου Ιρλανδίας θα λάβουν υπόψη τους το σωρευτικό αντίκτυπο σε αυτή τη φάση με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας είναι δύσκολο να διαπιστωθεί πραγματικά και να στοιχειοθετηθεί παραβίαση. Αν ο αναφερόμενος ωστόσο κατά τη διάρκεια της αναφοράς μας παράσχει επιπρόσθετες πληροφορίες, για παράδειγμα ότι δεν θα γίνει EIA για μία από τις εγκαταστάσεις ή ότι για παράδειγμα η μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου δεν λαμβάνει υπόψη τη σωρεστική δράση άλλων χιτά. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, ευχαρίστω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει την εξέταση του θέματο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ομιλίες τους και την ευέλικτη στάση τους. Πάντως, επί τη βάση αυτών που ακούσαμε, θεωρούμε ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η γνώμη την οποία εκφράζει ο αναφερόμενος διαφέρουν σε πολλά σημεία. Ορισμένα από τα σημεία αυτά λοιπόν παραμένουν ανοιχτά και ίσως θα χρειαστεί να δούμε αν η συλλογή περαιτέρω πληροφοριών ή μια αποστολή επιτόπου θα μπορούσε να βοηθήσει την κατάσταση. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Η κυρία Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλό θα είναι να έχουμε περαιτέρω ενημέρωση. Όπως είπαμε σήμερα το πρωί, σε αντίστοιχες περιπτώσεις, με αντίστοιχες αναφορές θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις λεγόμενες σορευτικούς παράγοντες, σορευτικούς δείκτες, γιατί είναι σαφές ότι τα κράτη-μέλη τείνουν να ιεραρχούν σε υψηλότερο βαθμό και επίπεδο τους οικονομικούς παράγοντες από ότι τους οικολογικούς. Η Επιτροπή Αναφορών λοιπόν θα πρέπει να παρακολουθήσει το θέμα από κοντά και εξακολουθεί να τρέχει σαν θέμα να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες από τις τοπικές αρχές. Κάποιες από τις πληροφορίες που έχουμε ζητήσει δεν έχουν δοθεί. Αυτά που μας είπε ο κύριος Λεόναρντ είναι πολύ σημαντικά. Μας είπε ότι στην περίπτωση της συγκεκριμένης μονάδας που λειτουργεί σήμερα οι κάτοικοι, οι περίοικοι έχουν πολύ κακές ε, εμπειρίες. Παρ' όλα αυτά η, η αντίστοιχη υπηρεσία περιβάλλοντος όχι μόνο θα επέτρεπε στη μονάδα αυτή να ανοίξει εκ νέου, όχι μόνο θα επέτρεπε να αυξήσει τον όγκο των σκουπιδιών τα οποία συλλέγει, και δεν είναι τυχαίο που την ημέρα πριν φτάσει για συζήτηση το θέμα εδώ άλλαξε η κυβέρνηση άποψη, η τοπική κυβέρνηση άποψη. Πάντως τώρα ζήτησαν κανονική άδεια αλλά δεν μας είπαν αν θα υπάρξει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αν θα ανταποκριθούν θετικά ή αρνητικά στο αίτημα για τη διεύρυνση της περιοχής και δεν έδωσαν και εξήγηση γιατί ε, έδωσαν άδεια να ανοίξει εκ νέου η μονάδα χωρίς να υπάρξει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αντίθετα από ό,τι θα έπρεπε να υπάρξει λόγω του μεγέθους μίλησα με κατοίκους της περιοχής και έχουν πράγματι υποφέρει. Είχαν πάρα πολλά προβλήματα, μολύνσεις, φλεγμονές στα μάτια, διάρειες, αλλεργίες, τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας δεν συμπεριλαμβάνουν τις λεγόμενους σωρευτικού παράγοντες. Και γι' αυτό το να περιορίσει κανείς την απάντηση στο ότι ανάλογα με το μέγεθος της εκμετάλλευσης ε, εξαρτάται και η περιβαλλοντική ή μη μελέτη επιπτώσεων, ε, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα περιοριστικό. Σας ευχαριστώ. Θα πρέπει να συνεχίσουμε νομίζω, δίνοντας το λόγο και σε άλλους συναδέλφους, για να θέσουν ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα απαντήσει η Επιτροπή. Κύριο Σταμπάζδη. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως με τη συνάδελφό μου κυρία Ντεμπρούν και θα ήθελα να κάνω μια γενική ερώτηση που με βασανίζει πάρα πολύ. Υπάρχουν οδηγίες για την αποτέφρωση των αποβλήτων και άλλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές λειτουργούν σωστά, εφαρμόζονται καλά ή όχι. Γιατί αυτό το πρόβλημα, αυτή η αναφορά που είναι πάρα πολύ θεμητή, καθώς και η επόμενη που είναι εξίσου θεμητή, δείχνουν ότι οι οδηγίες δεν βοηθούν στην πρόληψη καθόλου μάλιστα για τις ανητικές συνέπειες της προστασίας του περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό λοιπόν θα ήθελα να προτείνω, κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή μας, γιατί υπάρχουν πολλές αντίστοιχες καταστάσεις και πολλές αναφορές σχετικά, να το κοιτάξει σε συνεργασία με την Επιτροπή Περιβάλλοντος που είναι καθήλυνα αρμόδια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί διότι δεν υπάρχει εδώ καλή πρόληψη των ε, περιβαλλοντικών ζημιών και είναι μέγα πρόβλημα αυτό για μένα. και θα πούμε σε άλλους ότι δεν έχετε αρκετά ε, επιχειρήματα ή αρκετές αποδείξεις ότι γίνονται ζημίες. Εδώ δεν μπορούμε να αποδείξουμε όταν ε, σχεδιάζεται ένα έργο ότι θα κάνει ε, ζημιά στο περιβάλλον. Αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν προστατευμένες ζώνες φυσικά πάρκα, εθνική δρυμή κοντά σε μια πόλη. Αν δοθεί μια άδεια οικοδομική, αυτό σημαίνει ότι δεν λειτουργεί καλά η οδηγία προληπτικά. Πώς τους δίνουν άδεια. Υπάρχει λοιπόν αρκετή βάση για την πρόληψη των περιβαλλοντικών ζημιών. Αλλιώ δεν θα μπορέσει η δική μα Επιτροπή να ασχολείται με όλε αυτέ τι αναφορέ και να δίνει απαντήσει. θα πρέπει να παρακολουθήσουμε και αυτή την περίπτωση και άλλες, γιατί βλέπω μεγάλες αντιφάσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και στα Ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω αυτά που λέτε και έχετε δίκιο. Ενδεχομένως, εγώ δεν μπορώ να κρίνω. Απευθύνομαι στη γραμματεία και ρωτώ αν είναι αρμόδια η δική μας επιτροπή για αυτά τα θέματα. Για να θεώρησε οδηγιών ή για να κάνουμε τροπολογίες ή σχόλια. Στο παρελθόν το κοιτάξαμε αυτό, όπως είπε και ο κύριος Σταπάιτσι, και σε περιπτώσεις που πήγαν τα μέλη σε χωματερές επισκέψεις. Πολύ συχνά ε, η θέση που λαμβάναμε ήταν υπέρ των αναφερομένων. Στο παρελθόν λοιπόν τι διαπιστώσαμε σε τέτοιες περιπτώσεις και το λένε και αναφορές και εκθέσεις πεπραγμένων. δεν ορίζεται σαφώς η απόσταση μεταξύ ε, της κατοικημένης περιοχής και της χωματερής. Ε, το κοντά όμως πόσο είναι, να μην είναι πολύ κοντά. Ε, το κοντά πώς ορίζεται, ποιος ε, το ερμηνεύει. Αυτό ζητάει και ο κύριος Ταμπάιτζη. Υπάρχουν επιτροπές με νομοθετική αρμοδιότητα, που δεν είμαστε εμείς όμως, αλλά πολύ πιο φυσιολογικό είναι για μας, για την Επιτροπή και τη Γραμματεία, να έχουμε επαφές με τους ενδιαφερομένους, στη συγκεκριμένη περίπτωση τις αρχές της Βορείου Ιρλανδίας, τους ενδιαφερμένους στον κόσμο, για να ε, μας ενημερώνουν και να αντιδρούμε γρήγορα και να, να δείχνουμε ότι και ανησυχούμε και παρακολουθούμε όμως το θέμα. Τώρα θα δούμε, η Επιτροπή θα αποφασίσει, η Επιτροπή μας δηλαδή, τι συνέχεια θα δώσει σε αυτό. Ναι. Σημείωσα λοιπόν. Το ότι αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να ξεκινήσει τις επαφές με τις υπηρεσίες της ε, Βορείου Ιρλανδίας για να τις ε, ζητήσει και τη θέση τους. Θα το αναφέρω και στο τέλος. Άλλα σχόλια παρακαλώ για την συγκεκριμένη αναφορά. Αν όχι, να δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να απαντήσει στις ερωτήσεις που του τέθηκαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά το, την ερώτηση της κυρίας Δεμπρίν για το κατά πόσο οπότε χρειάζεται μάλλον ε, μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Σύμφωνα με το παράρτημα 1 της οδηγίας χρειάζεται τέτοια μελέτη σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις ε, απόρριψης αποβλήτων για την ε, αποτέφρωση χημικών αποβλήτων. Και εδώ μιλάμε για χιτά. Εδώ χρειάζεται τη δικασία screening όπου αναφέρεται όπου, υπάρχουν, όπου υπάρχει σημαντικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται ε, μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου και μεταξύ των κριτηρίων συγκαταλέγεται και το κριτήριο της ορευτικής δράσης. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι το κριτήριο αυτό θα πρέπει να λεφτεί υπόψη ε, από τις εθνικές αρχές όταν θα αποφασιστεί κατά πόσο οχητά συνεπάγεται σημαντικό αντίκτυπο ή όχι. Στα γαλλικά για τον κύριο Ταμπάιτζη, σε ό,τι αφορά την πρόληψη των κοινοτικών οδηγιών, εγώ έχω κάπως διαφορετική ερμηνεία. Θα έλεγα ότι η οδηγία 85337 αλλά και άλλες είναι κατεξοχή νομοθετικά εργαλεία με προληπτικό πνεύμα. Γιατί, Γιατί ε, ε, προβλέπουν μία διαδικασία αδειοδότησης πολλαπλών σταδίων ε, με δημόσια συμμετοχή και όλων των φορέων που ενημερώνονται εκ των προτέρων και μπορούν να επεμβαίνουν. Βεβαίω, για την οδηγία αυτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είμαστε απολύτω ικανοποιημένοι. Πρόσφατα δημοσίευσε μια έκθεση Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο για την εφαρμογή της οδηγίας και αρχές του έτους ε, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η οδηγία θα συζητηθεί σε σχέση με την ανάγκη αναθεώρησής της. Τώρα το θέμα ε, της ποιότητας των περιβαλλοντικών μελετών ε, ή της προληπτικής δράσης είναι πολύ σημαντικό και αν έχει να κάνει το Κοινοβούλιο ε, παρατηρήσεις εδώ με χαρά να τις χρησιμοποιήσουμε και να τις σημειώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στον αναφέροντα και να τον ευχαριστήσω εξ ονόματος όλων μας που παρευρέθηκε εδώ στην Επιτροπή μας και να ζητήσω να μας πει και τις εντυπώσεις του. Θεωρείτε ότι η συζήτηση αυτή συνέβαλε ή ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν και μελλοντικέ συζητήσει. Ευχαριστώ όλου σας για τα σχόλιά σας. Μας βοηθάει το γεγονός ότι ο κόσμος σε απόμαχρε περιοχέ στην Ιρλανδία μπορεί να υπολογίζει σε εσά. Έχει ήδη υπάρξει παραβίαση, θεωρεί η κοινότητα, όταν το 2006, όταν μια καταστροφική τέτοια εγκατάσταση που είχε ήδη κλείσει ξανά Και το γεγονός ότι δεν έγινε το 2006 μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου αποτελεί παραβίαση και αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί γιατί αυτό συζητιέται σε τοπικό επίπεδο επί σειρά μηνών γιατί δηλαδή, για ποιο λόγο δεν έγινε τέτοια μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Και θα ήθελα να το πω αυτό γιατί στην περίπτωση που θα είχε γίνει η μελέτη αντικτύπου θα είχε εξεταστεί, υπό... θα είχε εξεταστεί ο αντικτύπος όλων των χιτά μαζί και η ισορρευτική τους δράση. Επίσης θεωρώ ότι ένα από τα μεγάλα ζητήματα στην περίπτωση αυτή είναι ότι Μπορεί να λέμε ότι θα γίνει μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου, αλλά με ποια κριτήρια ε, γίνεται καταμέτρηση της ορευτικής δράσης στην περιοχή αυτή συμπεριλαμβανομένων όλων των εγκαταστάσεων, όλων των μονάδων. Ο Υπουργό δεν μου απάντησε τίποτα ουσιαστικά και σήμερα, αν ζητούσαμε να μας πούν συγκεκριμένα πώς γίνονται οι μετρήσεις, δεν νομίζω ότι θα λαμβάναμε απάντηση. Τα κριτήρια λοιπόν μέτρησης θα πρέπει να διευκρινιστούν και θα πρέπει να καταστούν ιδιαίτερως αντικειμενικά για να ξέρουν οι κοινότητες ότι είναι δίκαιη η μεταχείριση η οποία υπόκειται. Για να σας απαντήσω, Πρόεδρε, θεωρώ ότι ήταν καλή ακρόαση, ότι ήταν χρήσιμη συζήτηση, ότι γίνονται κάποια βήματα ε, προς μπροστά. Και ξέρω, είμαι πεπισμένος ότι αν συνεχιστούν οι έρευνε προς την κατεύθυνση αυτή, ο κόσμος στην κοινότητά μας θα είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη φορά, Πάλι από την Ιρλανδία. Του κυρίου David Rogers. Α, όχι. Υπήρξε μια μικρή αλλαγή. Δεν θα μιλήσει ο ίδιος ο αναφέρον, αλλά ο κύριος Κάσμαν που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν παρίσταται ο αναφέροντας. Γι' αυτό λοιπόν θα πάρει το λόγο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κ. Κάσμαν. Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως και στην προηγούμενη αναφορά και η αναφορά αυτή σχετίζεται με θέματα διαχείρισης χιτά στην Ιρλανδία στη Νότια Ιρλανδία αυτή τη φορά. Ο αναφέροντας εκφράζει τι ε, σοβαρές τους ε, ανησυχίες για τη ρήπανση του αέρα που προκύπτει από την λειτουργία του χιτά που βρίσκεται στο Καντιλάν στην βόρειο-ανατολική Ιρλανδία. Ο αναφέρον δηλώνει ότι δεν ε, τηρούνται σχετικοί όροι όπως και στην προηγούμενη φορά, η οδηγία για τους χιτά είναι η σχετική οδηγία και όπως αναφέρθηκε η οδηγία αυτή ορίζει λεπτομερείς όρους για να διασφαλίσετε η ασφαλής διαχείριση των χιτά προκειμένου να μην υπάρχουν περιβαλλοντικές ε, συνέπειες. Επικοινωνήσαμε με τις Ιρλανδικές Αρχές, οι οποίες και επιβεβαίωσαν ότι έχει έγκριση ο ΧΙΤΑ που λειτουργεί στην περιοχή αυτή. Η έγκριση είναι του 2003 και οι Ιρλανδικές αρχές επίσης επιβεβαίωσαν ότι υπήρξε μεγάλος αριθμός ενστάσεων και παραπώνων για διάφορα προβλήματα του ΧΙΤΑ τους πρώτους μήνες του 2007. Ο ΧΙΤΑ τον χιτάτε χειρίζονται οι τοπικές ε, αρχές, το Συμβούλιο της Κομιτείας εκεί. Και πρόκειται για μία υπηρεσία η οποία διαχειρίζεται τις ε, άδειες διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων και ε, εξασφαλίζει ότι τηρούνται όλοι οι σχετικοί όροι. Μετά από όλες τις ενστάσεις που υπέβαλαν οι κάτοικοι της περιοχής, η υπηρεσία ξεκίνησε σχετική έρευνα και όντως βρέθηκαν στοιχεία ανησυχητικά σχετικά με τον ΧΙΤΑ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις πρακτικές και τους ελέγχους και τη διαχείριση των αερίων του ΧΙΤΑ. Η υπηρεσία λοιπόν έκανε διάφορες επισκέψεις και εμπειρογνωμόνων για να εξεταστεί η επεξεργασία αερίου και κατέληξε σε συγκεκριμένες συστάσεις προς τις τοπικές αρχές. Οι Ιρλανδικές αρχές αναφέρουν ότι εφαρμόστηκαν οι συστάσεις αυτές που έγιναν και ότι θεωρούν ότι τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν μέσω της παρέμβασης του EPA, της, υπηρεσίας, ε, της περιβαλλοντικής υπηρεσίας. ενώ δηλαδή τις 7 οι ενστάσεις και τα παράπονα ήταν 18 του αριθμού, μετά ε, στο δεύτερο ήμιση ήταν μόλις 3. Και αυτό συνοψίζει την κατάσταση. Είναι σαφές ότι υπήρξαν προβλήματα κατά το πρώτο ήμιση του 2007 και οι εθνικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι υπήρξε παρέμβαση ότι ανέλαβαν συγκεκριμένες ε, δράσεις για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που είχαν καταγγελθεί. Έκτοτε δεν υπάρχουν πληροφορίες για συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία ενδεχομένως να ανακύπτουν ακόμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ. Θέλει κανείς να λάβει το λόγο για την αναφορά αυτή. όχι. Ωραία. Ολοκληρώνεται λοιπόν εδώ η συζήτηση για την αναφορά αυτή, μια που απουσιάζει και αναφερόμενος και δεν μπορούμε να κάνουμε ε, τίποτα παραπάνω. Παραμένει σε εκκρεμότητα αυτή η αναφορά. Θα ήθελα τώρα να έρθουμε στο επόμενο θέμα, που είναι από την πατρίδα μου, την Ουγγαρία. Η αναφορά αυτή, είναι παρόν αναφερόμενος. Έχετε λάβει το έγγραφο αυτό που έφερε μαζί του και μας ε, μοίρασε ο ενδιαφερόμενος. Ελπίζω να έχετε λάβει όλοι ένα αντίτυπο και θα παρακαλούσα τον κύριο Τίμπορ Τσάι, το δήμαρχο της πόλης Σεν Γκοτάρτ, να μας κάνει την παρουσίασή του. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ανάληψη των καθηγόντων σας και να σας ευχηθώ καλή τύχη. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω μερικές διαφάνειες για να συνοδεύσω την παρουσίασή μου. Tisztelt Bizottság, tisztelt Elnök Nagyon köszönöm, hogy Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι πάρα πολύ που ασχολούνται με τα προβλήματα τόσο αξιόλογοι άνθρωποι. Και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να μιλήσω εδώ ε, για την πόλη μου, το Σεν Κοτάρτ, το φυσικό δρυμό και το φυσικό ε, ε, πάρκο της περιοχής. Η πόλη Σεν Κοτάρτ είναι στο τριεθνές Αυστρίας, ε, Σλοβενίας, Ουγγαρίας. Απευθύνουμε μία έκκληση ε, σε βοήθεια και προς τους φίλους από την Αυστρία και τη Σλοβενία. Το Σεν Κοντάρτ είναι από τις 10 πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες τουριστικά είναι τουριστικός προορισμός και συνεργαζόμαστε και με τους Σλοβαίνους και με τους Αυστριακούς μας φίλους και γείτονες. Έχει γίνει μια επένδυση αποτέφρωσης εκεί ε, απορριμμάτων. Αλλά υπάρχουν κάποια προβλήματα, δύο-τρεις ε, παραβιάσεις. Είναι μια επένδυση κερδοσκοπική και καθόλου ε, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, διότι μεταφέρουν τα απόβλητα από απόσταση 500 χιλιόμετρων και πλέον για να αποτεφρωθούν στο εργοστάσιο αυτό. 350.000 τόνοι είναι η δυναμικότητα και μόνο το 1 δέκατο καλύπτεται. Οπότε δεν είναι θέμα δημοσίου συμφέροντος αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, διαπίστωσε ότι σε ό,τι αφορά την ατμοσφαιρική ρήπανση υπάρχουν αντιφάσεις ακόμα και στην παρασκευαστική φάση αυτής της μονάδας. Από τη μελέτη αντικτύπου που έγινε από τον Αυστριακό επενδυτή ε, ότι η εγκατάσταση αυτή υποτίθεται που είναι κοντά στα ουγγρικά σύνορα ε, ότι θα εκπέμπει ρήπαση μόνο προς την αυστριακή πλευρά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ούτε ανταποκρίνεται στις βέλτιστες ε, διαθέσιμες ε, τεχνικές. BAT όπως ονομάζεται αυτό. Ε, και παραβιάζει και τρεις βασικές οδηγίες της κοινοτική νομοθεσίας. και χρειάζεται αναθεώρηση ή ε, άδεια που εξέδωσε η Αυστρία. Εγώ δεν σας ζητώ τώρα να λάβετε μέρος σε μια διένεξη δύο γειτονικών πόλεων. Εμείς αγαπάμε πολύ την Αυστρία. Πηγαίνω με την οικογένειά μου διακοπές για σκι στην Αυστρία. Έχουν φανταστικό τουρισμό, πολύ ανεπτυγμένο. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνω Πώς είναι δυνατόν να το κάνουν αυτό σε μια περιφέρεια να εγκαθίσταται ένα τέτοιο εργοστάσιο χωρίς να ακούνε τους κατοίκους, τα δύο τρίτα των κατοίκων. 97% του πληθυσμού συμμετείχε σε δημοψήφισμα στο Σεν Κοντάρτ και απέρριψαν οι κάτοικοι ε, την εγκατάσταση αυτού του εργοστασίου εκεί. Και είναι και προηγούμενο αυτό, μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο στην Ευρώπη. Μιλούμε για την Ευρώπη των περιφερειών. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια προβλήματα άλλη απαράδεκτα. Δεν μπορεί η περιφέρεια να μην έχει λόγο ε, για μια επένδυση που γίνεται στα 500 μέτρα από τα σύνορά μας. Ε, σίγουρα χρειάζεται να θεώρησε αυτή η ρύθμιση. Ακούσαμε τα θέματα της προηγούμενης αναφοράς και θα ήθελα να το επιβεβαιώσω κι εγώ και να σας ε, ζητήσω ή να σας ρωτήσω ε, πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε. Καλές οι άδειε και η προετοιμασία, αλλά δεν θα πρέπει να ρωτούμε και τους γείτονε. Εδώ είμαστε στον 21ο αιώνα, δεν μπορούμε να έχουμε μεθόδους του 20ου για να μην πω του 19ου. Παρακαλώ να ε, αναθεωρηθεί αυτή η περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας, λέει η Πρόεδρος. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρακαλώ. Thank you, Mrs. So, the commission for this petition... Η Επιτροπή για την αναφορά αυτή έχει αποστείλει ήδη λεπτομερή ανακοίνωση που αναφέρεται σε όλες τις οδηγίες στις οποίες γίνεται αναφορά στην αναφορά για την παραβίαση της οδηγίας για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, για τους οικοτόπους, για την αποτέφρωση ε, αποβλήτων, IPCC, και στην ανακοίνωση έχουν αναφερθεί οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εν συντομία, λοιπόν, αναφερθώ στα σημεία τα οποία ανέφερε και ο αναφέροντας. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την ποιότητα του περιβαλλοντικού αντικτύπου, της μελέτης περιβαλλοντικού αντικτύπου, δυστυχώς η σχετική οδηγία δεν θέτει ποιοτικά πρότυπα. Και λέμε συχνά ότι ακόμα και από σε αποβλήτων ουσιαστικά μπορεί να δημιουργηθεί, να κατασκευαστεί στον Άγιο Πέτρο της Ρώμης βάσει της οδηγίας. Από τη στιγμή που έχει γίνει η μελέτη αντικτύπου και έχει εκφραστεί η γνώμη του κοινού, θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να αποφασίσουν. Γι' αυτό λοιπόν το δεύτερο επιχείρημα για την διαβούλευση του κοινού που ανέφερε ο ενδιαφερόμενος δεν ισχύει γιατί πρόκειται ουσιαστικά μόνο για τη μία διαβούλευση με το κοινό. Την απόφαση τελικά τη λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές οι διαβουλεύσει δεν είναι δεσμευτικέ και να τονίσω ότι υπάρχουν και παρόμοια προβλήματα σε άλλες περιοχέ της Ένωσης, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά κατασκευή τέτοιων ε, εγκαταστάσεων. Επίσης, αναφέρονται οι καλύτερε διαθέσιμες τεχνολογίες, τις οποίες θέτει ως όρο η οδηγία IPCC. Πρόκειται για κάποια έγγραφα κατευθυντήρια, αν θέλετε, τα οποία έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία όμως ακριβώς αποτελούν απλά κατευθυντήρια έγγραφα και τίποτα παραπάνω. Χρησιμοποιείτε μία από τις τεχνολογίες που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. Μπορεί όχι η καλύτερη, αλλά μία από αυτές που αναφέρονται. Τέλο αναφέρεται η αρχή τη εγκύτητα και η παραβίαση αυτή που αναφέρεται στην οδηγία πλαίσιο. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η μέθοδος επεξεργασίας των αποβλήτων. Πριν μιλούσαμε για χιτά, τώρα μιλάμε για αποτέφρωση αποβλήτων. Η Κομισιόν θεωρεί ότι η αποτέφρωση ε, αποβλήτων είναι καλύτερη από την υγειονομική ταφίτη τους από περιβαλλοντική άποψη. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί, να στοιχειοθετηθεί η παραβίαση της αρχής της εγκύτητας. Συνοψίζοντας πρέπει να πω ότι με τις πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε παραβίαση. Εφόσον μας δοθούν καινούργιε πληροφορίες, ευχαρίστω να ξανακοιτάξουμε την αναφορά. Και εξ όσων καταλάβαμε, η άδεια που ζητήθηκε και χορηγήθηκε δόθηκε υποεθνική δικαιοδοσία γιατί όπως ξέρετε τα εθνικά δικαστήρια είναι κοινωτικά δικαστήρια. Σας ευχαριστώ. Έχουν ζητήσει κάποιοι συνάδελφοι το λόγο. Ο κύριο Άντερ έχει πρώτο ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής, Εσχολούμαι με τα θέματα της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Και έχουμε πάρα πολλά θέματα τα οποία συζητάμε εκεί, τα οποία είναι ανάλογα με αυτά που συζητάτε εδώ. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα να ζητήσω την υποστήριξή σας για την πρωτοβουλία του Τσέντ Κοτάρντ. Νομίζω ότι αυτή η επένδυση είναι μια κακή επένδυση οι κάτοικοι της περιοχής έχουν δίκιο, οι περίοικοι έχουν δίκιο. Η προστασία του περιβάλλοντος, η συνεργασία ανάμεσα στις περιφέρειες, η προστασία γενικότερα των περιοχών αυτών είναι λόγια τα οποία ακούμε σε καθημερινή βάση. Μιλάμε για μια περιοχή στην οποία κατοικούν Ούγγροι, Σλοβαίνοι, Αυστριακοί και προσπαθούν να παρουσιάσουν τις περιοχές αυτές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να δώσουν την καλύτερη εικόνα. Όπως είπε ο δήμαρχος του Τσεντ Γκόταρντ, στην περιοχή υπάρχουν εθνικά πάρκα. Αυστριακοί, Ούγγροι και Σλοβαίνοι διαμαρτύρονται από κοινού εναντίον αυτής της οικονομικής προσπάθειας. Ο Δήμαρχος και αυτός εκφράστηκε αντίθετα είπε ποιες είναι οι προσπάθειες της περιοχές να αναπτυχθεί, η αματικός τουρισμός, είδατε φωτογραφίες, γίνεται μία προσπάθεια. Και αυτό δεν αφορά μόνο το Τσεντ Γκόταρντ αλλά και άλλες περιοχές και μάλιστα και σε γειτονικές χώρες οι οποίες επωφελούνται από την προσπάθεια αυτή. Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό το οποίο ήδη ακούστηκε. Υπάρχει μια προσπάθεια που γίνεται στην συγκεκριμένο χώρο για να οικοδομηθεί, για να κατασκευαστεί μια μονάδα καύσης η οποία θα έχει την δυνατότητα να απορροφά δεκαπλάσιες ποσότητες απορριμμάτων από αυτά τα οποία παράγει το Burgenland. και όμως η επένδυση αφορά 10 φορές το δυναμικό παραγωγής απορριμμάτων. Θα έπρεπε να ε, κατασκευαστεί σε άλλη περιοχή πάρα πολύ κοντά στο Γκράτς αυτή η μονάδα. Αλλά οι πολίτες οι Αυστριακοί διαμαρτυρήθηκαν και τώρα ξαφνικά αποφασίστηκε να έρθει στο Τσεν Κόταρντ. Προφανώς και θα πρέπει να υπάρξει φροντίδα για τα απόβλητα, για τα απορρίμματα, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Υπάρχει επίσης μια, ένας τρίτος αστριακός δήμος που συμφωνεί να γίνει μια τέτοια μονάδα καύσης στο Λίντς. Οπότε γιατί επιμένουν να κατασκευάσουν τη μονάδα αυτή σε μια περιφέρεια όπου όλοι οι περίοικοι διαμαρτύρονται και όχι σε άλλες περιφέρειες όπου οι δημοτικές αρχές έχουν ήδη εκδώσει άδειε οικοδόμησης της μονάδας καύσης. Αυτές οι μονάδες θα μπορούσαν να φροντίσουν και τα απόβλητα τα οποία παράγονται στην περιοχή του Μποργενλάντ. Υπάρχουν και κάποια νέα στοιχεία λοιπόν τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα οποία ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακούσαμε διάφορα και για τις κλιματολογικές αλλαγές. Οι κάτοικοι της περιοχής έζησαν τις αλλαγές αυτές στο πετσί τους. Φέτος ξεχύλισε ο ποταμός Ραμπ τρεις φορές. Έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ ύψους ο ποταμός αυτός. Και αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις κοιλάδες γύρω από τον ποταμό Ραμπ φέτος λίγα ε, εκατοστόμετρα έλειψαν για να μην ξεχυλήσουν και τα δύο αποδοχής των ποταμών αυτών και οι πλημμύρες αποκτήσουν διαφορετικές διαστάσεις. Λοιπόν, τι είδους ζημιές οικολογικές θα δημιουργηθούν στο μέλλον, πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Οφείλουν λοιπόν τα μέλη αυτής της Επιτροπής όταν παίρνουν αποφάσεις γύρω από τα θέματα αυτά να μην αγνοούν τα εξή. Μια τέτοια μονάδα καύσης, μια τέτοια κάμινος μπορεί να οικοδομείται ε, στα σύνορα εθνικών πάρκων. Μια τέτοια μονάδα. να καταστρέψει την προσπάθεια συνεργασίας τριών χωρών και τριών περιοχών μεθοριακών. Δεν θα πρέπει να γίνεται αυτό. Και τέλος θα πρέπει να αγνοήσουμε τις διαμαρτυρίες των Ούγγρων, των Αυστριακών και των Σλοβαίνων πολιτών. Αυτή η μονάδα καύσης θυμίζω ότι θα χτιστεί και με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιλάμε για 130 εκατομμύρια ευρώ. Και τέλος η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να διακινδυνεύσει μια τόσο μεγάλη επένδυση να οικοδομηθεί σε μια περιοχή η οποία ε, κινδυνεύει και από τις πλημμύρες σε υψηλό βαθμό. Αυτό που καταλαβαίνετε ότι θα προκαλούσε πολύ πιο σημαντικές ζημιές από αυτές που έχουμε προβλέψει μέχρι τώρα. Έχουμε ακούσει ότι μία κάμινος θα μπορούσε να χτιστεί και κοντά στη βασιλική του Αγίου Πέτρου. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει. Κανένας δεν θέλει να βλέπει την καμινάδα μιας τέτοιας μονάδας. και αυτό δεν θέλουν να δούνε και στο σπίτι τους και δίπλα από τις δικές τους εκκλησίες οι κάτοικοι του Τσεντ Κόταρντ. Η λύση είναι στα χέρια των Αυστριακών αρχών. Ο άλλος χώρος στον οποίο δεν θα υπάρχουν προβλήματα είναι 80 χιλιόμετρα μακριά. Σιγά την απόσταση. Ευχαριστώ κύριο Τσάμπα Ταμπάιντε. Κυρία Πρόεδρε, η αναφορά αυτή είναι πάρα πολύ θεμητή και αιτιολογημένη. Είναι σαφές και υπάρχουν πολλές αντιστοιχίες και ομοιότητες με άλλες αναφορές που εξετάσαμε στο παρελθόν και προηγουμένως. Μου είπε κάτι πολύ σημαντικό ο κύριος Λόου και ερωτώ αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα στη γραμματεία να γίνει ένα συμπίλημα, μία σύνοψη της βαρθούς εμπειρίας της Επιτροπής Αναφορών για να τη στείλουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος που είμαι και εκεί μέλος, αναπληρωματικό όμως. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος επαναλαμβάνω για να κάνω ό,τι μπορώ μαζί με τους συναδέλφους μου γιατί είναι σαφές και συμφωνώ απολύτω με τον κύριο Λόου υπάρχουν προβλήματα με τις οδηγίες αυτές σε ό,τι αφορά την απόσταση. Διότι αν οι οδηγίες αυτές δεν, πώς να το πω, διευκρινίζουν ότι στις προστατευμένες περιοχές της Natura 2000 ή σε πόλεις όπως είναι το Σεν Κότατ αν δεν προσδιορίζεται σε πόσα χιλιόμετρα απόσταση μπορεί να κατασταθεί ένα τέτοιο εργοστάσιο ε, τότε αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και δεν είναι το πρόβλημα της Ουγγαρίας αυτό μόνο. Και ο συνάδελφος κύριος Άντερ το ξεκαθάρισε πολύ καλά. Δεν είναι ουγγρικό το πρόβλημα, είναι τριευθές. Και πολύ περισσότερο υπάρχει και μια άλλη διάσταση του προβλήματος. Ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να μεταφέρει τη ρήπανση εντό εισαγωγικών σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να την εξάγει και πολύ περισσότερο μπορεί να ρηπαίνει μια προστατεμένη περιοχή, τη δική του προστατευμένη περιοχή. Διότι το Εθνικό Πάρκο Ράτζα είναι στην Αυστρία και αυτό απειλείται. Λοιπόν, αφορά και τις τρεις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό και ακόμα και η οικονομική άδεια ε, είναι πρόκληση που δώσανε να χτιστεί εκεί το εργοστάσιο. Αυτό και μόνο είναι παραβίαση της προστασίας του περιβάλλοντος στην Ευρώπη γενικώ. Και αυτό αποδεικνύει την έλλειψη καλής βούλησης. Γι' αυτό χρειάζεται αναθεώρηση. Και έχω ένα μικρό ζήτημα με εσάς κύριε εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διότι η οδηγία για την ατμοσφαιρική ρήπανση λέγει ότι θα πρέπει να καταβάλλονται οι πληρωμές και αποζημιώσεις μετά από την παραβίαση, είπαμε, αφού διαπιστωθεί η παράβαση. Πρόληψη καμία. Οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Αν διαβάσετε την τελευταία φράση στο ε, φάκελό μας, θα δείτε ότι καταβάλλονται οι πληρωμέ και αποζημιώσεις εφόσον εγκατασταθεί το εργοστάσιο κατόπιν εορτή. Πού είναι η πρόληψη στι οδηγίε μα, δεν υπάρχει καμία πρόληψη. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει οπωσδήποτε να αναθεωρηθούν κάποιε οδηγίε να δούμε ποιε αφορούν την προστασία του περιβάλλοντο προ όφελο όλων των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε και να βρούμε μια λύση, διότι εάν χτιστεί αυτό το εργοστάσιο, χαιρετίσματα. Ε, θα είναι ήδη πολύ αργά. Θα έχουν γίνει ζημίες και ο κύριος Άντερ πρόσθεσε και κάτι ακόμα, ότι υπάρχει και μια άλλη απειλή από ε, τις πλημμύρες. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθήσουμε το θέμα αυτό και να βρούμε μια λύση από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Igen, ευχαριστώ. Ο äh, Λαμβάνουμε όλο και πιο πολλές ε, αναφορές που έχουν να κάνουν με τη σχέση μεταξύ των κρατών μελών. Και θα ήθελα να συμφωνήσω με τον προηγούμενο μιλητή στο σημείο αυτό και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην δημιουργηθούν εντυπώσει ότι εσκεμμένα κάποιες χώρες ε, μεταφέρουν τις εγκαταστάσεις αυτές στα σύνορά τους για να τις φορτώσουν στους γείτονες. Γιατί στο εσωτερικό τους τα κράτη-μέλη έχουν πολύ ακριβείς και αυστηρούς κανόνες και για παράδειγμα στη Γερμανία ισχύουν πολύ αυστηροί κανόνες. Για παράδειγμα, αν ε, χτίσουμε μια τέτοια μονάδα είναι πολύ σαφείς οι κανόνε για το πόση απόσταση θα πρέπει να τηρήσει από το γείτονα. Στα μπαλκόνια, για παράδειγμα. Άρα θα πρέπει να διατυπωθούν μεγαλύτερη ακρίβεια οι προδιαγραφές αυτές και για τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών και έχετε δίκιο. Αν είναι πρώτα να χτιστεί η εγκατάσταση και μετά να συνεργαστούν ε, τα κράτη-μέλη, χαίρο πολύ. Αν υπάρχει κάποιο έλλειμμα, θα πρέπει να το ορίσουμε εξ αρχής. Και θεωρώ ότι είναι μεγάλη, μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό παρουσιάζεται και σε άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου κατασκευάζονται για παράδειγμα αναμογεννήτριες και δεν συμφωνεί το ομοροκράτος. Νομίζω λοιπόν ότι ως Επιτροπή θα πρέπει να το διαπιστώσουμε αυτό, ότι υπάρχει στο σημείο αυτό πρόβλημα και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εξή. Αν ε, όντω πρόκειται για περιοχή που πλήττεται από πλημμύρε, γιατί και εγώ από τη Σαξονία είμαι, που έχουμε τεράστια προβλήματα και μπορεί επί 20 χρόνια να μην είχαμε προβλήματα, αλλά μετά από 20 ολόκληρα, προβλή... Ε, μετά από 20 ολόκληρα χρόνια που δεν υπήρχε πρόβλημα, παρουσιάστηκαν και πάλι προβλήματα. Άρα ε, θα πρέπει να κοιτάξουμε όντω, να μην κατασκευάζονται τέτοια έργα σε περιοχές που πλήττονται από πλημμύρες. Αν θα μπορούσε λοιπόν να μου απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ρωτήσω και στην Αυστρία τι γίνεται και επίσης ε, για την προστασία από πλημμύρε υπάρχουν και σχετικέ νομικέ προδιαγραφέ. Αυτά τα δύο προβλήματα θεωρώ ότι υπάρχουν σε σχέση με την ε, αναφορά. Η κυρία Ντεμπρούν, ευχαριστώ. Να κάνω ένα μικρό σύντομο σχόλιο. σε σχέση με ένα από τα θέματα τα οποία ανέκυψαν και προηγουμένως. Το θέμα της μελέτης περιβαλλοντικού αντικτύπου και της ορευτικής δράσης. Το θέμα δεν είναι μόνο αν γίνεται μελέτη. Το θέμα είναι και πώς γίνεται η μελέτη, τι ποιότητα μελέτης έχουμε, αν το κράτος μέλος ξέρει ποια κριτήρια ισχύουν και πώς θα πρέπει να εφαρμοστούν στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται αναφορικά και με τη σωρευτική δράση. Αυτό έχει ήδη έχει ανακύψει τρεις φορές σήμερα. Έχουμε ακούσει το ίδιο στοιχείο σε τρεις διαφορετικές αναφορές. Και αυτή η σημερινή μελέτη που είχαμε σήμερα το πρωί. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό ως Επιτροπή να εξετάσουμε το θέμα αυτό και να ζητήσουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το λάβει υπόψη στις συζητήσεις με τα κράτη-μέλη. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν έχετε άλλο τίποτα να πείτε για αυτή την αναφορά, θα ήθελα να συνοψίσω λίγο τη συζήτηση, γιατί ήταν λίγο μακροσκελής. Χαίρομαι που βλέπω τέτοια επίδειξη αλληλεγγύης και σύμπνοιας σε σχέση με την αναφορά αυτή. Και, γιατί μίλησαν και συνεισέφεραν και κάποιοι συναδέλφοι που δεν θίγονται άμεσα. Και πέρα από πολιτικές ομάδες ε, οι παρατάξεις. Συμφωνούμε λοιπόν, αυτό δεν ε, γνωρίζει κομματικά σύνορα το θέμα. Ε, τα ζητήματα περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντικά. Επίσης, έχω την αίσθηση ότι υπήρξε ένα αίτημα προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις αναφορές από την ε, Ιρλανδία και την Ουγγαρία, το Σαν Γκόταρτ. Στην αρχή ε, τη της συνεδρίασής μας ακούσαμε μια παρουσίαση για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Αλλά κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και προστατευμένοι. Δηλαδή, όταν ε, υφίστανται τις συνέπειες μια ανετικής ε, απόφασης, θα πρέπει να νιώθουν ασφαλείς ότι δεν θα χαθούν στους δεδάλους ε, της νομοθεσίας και της γραφειοκρατίας. Η αλήθεια θα πρέπει να θειαδεύσει και να είναι πιο ισχυρή από τη γραφειοκρατία. Με κάθε σεβασμό το λέω αυτό προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το πω. Ακούσαμε πολλά επιχειρήματα υπέρ και κατά και νέα στοιχεία έχουν ανακύψει σε αντίθεση με άλλες αναφορές. Μίλησαν και ο κύριος Άντερ και ο αναφερόμενος και για τον κίνδυνο πλημμυρών. Αυτό το νέο λοιπόν στοιχείο νομίζω μας υποχρεώνει να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή, να τη διατηρήσουμε στη μέση διάταξη και θα παρακαλούσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει το θέμα. Και τέλος, να πούμε και κάτι θετικό στον αναφερόμενο. Ο επικεφαλής της γραμματείας με ενημερώνει ότι ελήφθη απόφαση ε, στην Επιτροπή Αναφορών να σταλεί επιστολή προς την Αυστριακή κυβέρνηση όταν θα το αποφασίσει η Επιτροπή μας. Και θα παρακαλούσα την Επιτροπή να εγκρίνει την πρόταση αυτή. Για να αποστείλουμε λοιπόν μια επιστολή προς την κυβέρνηση της Αυστρίας και να λάβει σοβαρά υπόψη την αντίσταση του ουγγρικού πληθυσμού. Ευχαριστώ πολύ και το Δήμαρχο. Τελευταία αναφορά τώρα ε, στο κεφάλαιο του περιβάλλοντος. Ο κύριος Γιαρέχο και άλλη παράκληση. Ε, θέλει αρμόδια επιτροπή, θα πρέπει να λάβει και αυτή η επιστολή. Γιατί με ενδιαφέρει πως έχει η ενόμη ε, σε περίπτωση οικοδομικών ε, αδειών και κατασκευών και οικοδομών σε παραμεθόριες περιοχές. Τι συμβαίνει εκεί, γιατί έχουμε όλη την εντύπωση ότι δεν συνεννοούνται αρκετά οι χώρες μεταξύ τους και εκεί χρειάζεται μάλλον νομοθετική ρύθμιση. Εμείς όμως δεν είμαστε αρμόδια Επιτροπή επί της ουσίας, αλλά ε, θα πρέπει να το διαβιβάσουμε σε άλλη Επιτροπή για να ασχοληθεί καλύτερα με το θέμα και πιο αρμόδια από μας. Η Πρόεδρος. Ναι, σημαντικό αυτό το σχόλιο. Υπάρχει δυνατότητα πράγματι να δώσουμε συνέχεια. Τώρα, τελευταία αναφορά για το περιβάλλον. Αλλά νομίζω που σιάζει ο αναφερόμενος η ε, αναφερόμενη μάλλον, η κυρία Βερόνη Καντίνη. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομο. Πρόκειται για τη γραμμή των τρόλεϊ της Μπολόνια. Το δίκτυο ΣΥΒΙΣ. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει γίνει δεν είναι η σωστή ή δεν έχει γίνει με σωστό τρόπο. Ο αναφερόμενος θεωρεί ότι η έκθεση η οποία έχει παρουσιαστεί πρέπει να ενημερωθεί. Εμείς δεν ακολουθούμε το επιχείρημα αυτό, γιατί η οδηγία δίνει την δυνατότητα στα κράτη-μέλη μεγάλη διακριτική ευχέρεια σχετικά με την αξιολόγηση ε, κάποιων προγραμμάτων και για το αν θα πρέπει να ενημερώνονται οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν βλέπουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση παραβίαση της οδηγίας γιατί δεν είναι δυνατόν να αποδείξουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν υπερβάλλει στη συγκεκριμένη περίπτωση οι Ιταλικές αρχές. Δεν έχουμε στοιχεία δηλαδή και δεν μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε ε, κάποια στοιχεία παραβίασης της οδηγίας για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ευχαριστώ. Δεν μπορούμε λοιπόν να δώσουμε συνέχεια στη συγκεκριμένη οδηγία. Θα την κλείσουμε λοιπόν και θα περάσουμε στην επόμενη ομάδα αναφορών για την αναγνώριση πτυχίων και δεξιοτήτων. Η πρώτη αφορά μια γαλίδα αναφερμένη. Αλλά δεν είναι παρούσα. Δεν το ήξερα. Οπότε για μια ακόμη φορά ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα λάβει το λόγο. Η κυρία Σράιερ. Πρόκειται για τη λήψη υπόψη της επαγγελματικής εμπειρίας που εργάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατά πόσον πρέπει να ληφθεί υπόψη στην τοποθέτησή της στο δημόσιο τομέα της Γαλλίας η εμπειρία η επαγγελματική που έχει αποκτηθεί σε άλλο κράτος μέλος θα λαμβάνεται υπόψη για την πρόσβαση στον δημόσιο τομέα της συγκεκριμένης χώρας και θα λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία και η προϋπηρεσία όπως εφαρμόζεται στους ίδιους τους πολίτες στην ίδια χώρα. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία επιπαραβάση εναντίον της Γαλλίας. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας οι γαλλικές αρχές υιοθέτησαν καινούριου κανόνες για τον δημόσιο τομέα. Μετά την υιοθέτηση αυτών των μέτρων, πιστεύουμε ότι θα βρίσκονται λύσεις σε τέτοιου είδους προβλήματα συμβατές με τα κοινοτικά μέσα και γι' αυτό σταμάτησε η διαδικασία προσφυγής επί παραλήψης. Στα πλαίσια αυτά, οι γαλλικές αρχές δημιούργησαν την λεγόμενη Επιτροπή Ισοτιμιών, Commission de όπου όλοι που έχουν αποκτήσει επαγγελματικές ε, ε, εμπειρίες σε άλλες χώρες αξιολογούνται. Η περίπτωση αυτή αξιολογήθηκε τον Οκτώβριο του 2007 αλλά οι πληροφορίες δόθηκαν στον αναφερόμενο μόνο ένα χρόνο μετά. Δεν ελήφθη υπόψη η επαγγελματική εμπειρία γιατί είχε διακόψει τη σταδιοδρομία της που κράτησε ε, περισσότερο από όσο επιτρέπεται στο γαλλικό νόμο. Θεωρούμε ότι ο όρος της συνέχειας σε μια εργασιακή σχέση είναι έμεση μορφή διάκρισης. Η μετακίνηση ενός εργαζομένου σε άλλη χώρα δεν πρέπει να οδηγεί στον σεβασμό του γαλλικού νόμου ε, ο οποίος ε, λέγει, προβλέπει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει διακοπή μεγαλύτερη από τρίμηνη στη συνεχή επαγγελματική δραστηριότητα. Ζητήσαμε την άποψη των γαλλικών αρχών και μας ενημόρισαν ότι με ένα νέο διάταγμα του Απριλίου του 2009 έχει αλλάξει και ο όρος της συνέχειας δεν υπάρχει πλέον. Οι αρχές τώρα της Κομισιόν θα έρθουν σε επαφή με τις γαλλικές αρχές για να δούμε ακριβώς τι θα συμβεί με τον αναφερόμενο, με την αναφερομένη και θα σας ενημερώσουμε όταν έχουμε νέα στοιχεία. Ευχαριστώ. Κύριε Σλάου, μια ερώτηση γιατί ήταν από τις πρώτες αναφορές που ε, ε, πήρα στα χέρια μου όταν ήρθα στη γραμματεία και κρεμεί εδώ και καιρό. Και επανειλημμένα μας είχαν διαβεβαιώσει ότι οι γαλλικές αρχές επιλαμβάνονται. Ε, ε, η αναφερμένη όμως έρχεται ξανά και ξανά και μας λέει ότι δεν λύνεται. Ε, Πόσο καιρό χρειάζεται η επαλήθευση και η επιβεβαίωση, εν πάση και πότε θα τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Για τη Γαλλία είχαμε πάρα πολλά παράπονα και καταγγελίες και ξεκινούμε ε, προσφυγή επί παραβάση κατά της Γαλλίας έχει φτάσει στο δικαστήριο. Είπαμε ότι εισήστησαν αυτή την Επιτροπή Ισοτιμιών, Κομισιόν και ε, αναθεωρούνται όλες οι περιπτώσεις και μόλις τον περασμένο Οκτώβριο ενημερώθηκε η αναφερομένη για τη τελική έκβαση. Και όταν ε, ε, ρωτήσαμε και εμείς τι γίνεται, φάνηκε ότι υπάρχουν επιπλέον κανόνες που αφορούν το συγκεκριμένο κλάδο εργαζομένων. Επιπλέον προϋποθέσεις. Στη Γαλλία, όπως ξέρετε, υπάρχουν 1.600 κατηγορίες εργαζομένων με ειδικούς κανόνες. Φτιάχνουν κάποιους κανόνες ε, πλαίσιο που διέπουν τη λειτουργία της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ε, αυτών των σωμάτων, ας πούμε, εργαζομένων, Και δεν ε, λαμβάνεται υπόψη στη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων αυτή η επαγγελματική εμπειρία. Το γενικό πρόβλημα έχει λυθεί με την έγκριση νέων κανόνων, τώρα τα επιμέρους. Ευχαριστώ. Ε, ε, κυρία Γκουρίνη, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, όντω είναι μια δυσκολία αυτή τη στιγμή στην Αλία για την αναγνώριση των διπλωμάτων και της επαγγελματικής εμπειρίας και δεν μιλούμε για εξωτερικό, μιλούμε για χώρες Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να αλλάξει αυτό. Το γνωρίζω. Εγώ έκανα διαβήματα στην κυβέρνηση. Υπάρχει βούληση στην κυβέρνηση για πλήρη αναγνώριση. Αντίθετα, η διοίκηση είναι πάρα πολύ αργή και έχουμε ολιγορίες, θα πρέπει να επιμείνουμε, διότι αυτό είναι παράλογο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κανονικά. Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να σπουδάζει, να εργάζεται, να κάνει άσκηση stage παντού. Και αυτό είναι και μία από τις ε, θετικές πτυχές και ισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον. Είπατε ότι υπάρχουν ειδικοί κανόνες στα δικαστήρια. Όχι, δεν είναι ειδικοί κανόνες στα δικαστήρια. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει νομολογία, ο κανόνας είναι ίδιος παντού. Από εκεί και πέρα η ερμηνεία του νόμου μπορεί να είναι διαφορετική. Αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει όλοι μαζί να προχωρούμε από κοινού. Για τους νέους είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να μπορούν να δικινούνται ελεύθεροι εργαζόμενοι. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι το πρόβλημα αυτό, η αρχή της συνέχειας καταργήθηκε η προϋπόθεση αυτή. Θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη στη συγκεκριμένη περίπτωση της αναφερμένης αυτής. Είναι νέο το ζήτημα αυτό που έχει ανακύψει και έχει διορθωθεί στους κανόνες. Δεν ξέρω. Δεν είπα τίποτα για δικαστήριο εγώ. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε και την συζήτηση για αυτή την αναφορά. Η επόμενη αναφορά, σε παρόμοιο, στον ίδιο κλάδο, δεν παρίσταται ο αναφέρον. Γι' αυτό λοιπόν να ζητήσω από την Επιτροπή. Μιλάμε για τα διπλώματα στη Γερμανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η γερμανική νομοθεσία για την αναγνώραση των πτυχίων αυτών δεν συμβαδίζει με το κοινωτικό δίκαιο. Γι' αυτό λοιπόν το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σχετικό έγγραφο προς τη Γερμανία ζητώντας να αλλάξει ο νόμος αυτός, να τροποποιηθεί προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση της γερμανικής νομοθεσίας με το κοινωτικό δίκαιο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις διατάξεις επαγγελματικών προσόντων και τη σχετική οδηγία. Τον Ιούνιο του 2009 που έγινε η τελευταία ε, αναφορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι γερμανικές αρχές πλέον μας έχουν ενημερώσει ότι έχει τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία και ότι συμμορφώνεται πλέον με το τεχνητικό δίκαιο. Εκρεμή και δικαστική ε, υπόθεση στο γερμανικό ε, δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει την, ε, τι θα αποφανθεί το δικαστήριο, γιατί μόνο τα εθνικά δικαστήρια είναι αρμόδια σε πρώτη φάση για να εξασφαλίσουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων του αναφερόμενου. Σε ό,τι αφορά δηλαδή την αναγνώριση του πτυχίου του αναφέροντα. Περιμένουμε λοιπόν την απόφαση του δικαστηρίου. Αν είναι υπέρ του αναφέροντα, η Επιτροπή σκοπεύει να κλείσει την υπόθεση αυτή. Αν η απόφαση του δικαστηρίου είναι κατά του αναφέροντα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσον λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις της σχετικής οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα. Και σε περίπτωση που αποφανθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν πληρούνται οι σχετικοί όροι, θα προσέχουμε την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο 10. Θα σας κρατήσουμε ενημέρους για τις εξελίξεις στην υπόθεση αυτή. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε για την απάντηση αυτή. Και έχουμε τώρα μία μαλτέζικη αναφορά και πάλι δεν είναι παρόν ο αναφέροντας. Να ζητήσω λοιπόν να σχολιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Αμπέλα ο αναφέροντας ε, ζητά να αναγνωριστεί ε, τα πτυχία του ως ε, μηχανικός στη Μάλτα. Η Μάλτα αποφάσισε ότι υπήρξε παραβίαση από πλευράς των μαλτεζικών αρχών γιατί σε πρώτη φάση αγνώρισαν πλήρως τα προσόντα του αναφέροντα και κατά δεύτερον δεν του έδωσαν την επιλογή μεταξύ των δύο μέτρων που προβλέπονται από την οδηγία, είτε δηλαδή μια περίοδο προσαρμογής, είτε ε, μια εξέταση. Τους τελευταίους τρεις μήνες παρουσιάστηκαν τέσσερα περιστατικά, τα οποία ε, κάνουν την Επιτροπή να πιστεύει ότι πλέον η Μάλτα πληρεί τον, την ε, Οδηγία 36 του 2005. Καταρχάς, ε, ο αναφέροντας μας ανέφερε μέσω email ότι όντως έλαβε πλέον την ε, επιλογή μεταξύ των δύο μέτρων και στις 19 Ιουνίου ο αναφέροντας αποφάσισε να ακολουθήσει την οδό της περίοδου προσαρμογής. 24 Ιουνίου της ε, βιντεοδιάσκεψη του Συμβουλίου Μηχανικών και των Μαλτεζικών Αρχών επιβεβαιώθηκε ότι όντως θα πρέπει να δοθεί αυτή η επιλογή στον αναφέροντα μεταξύ των διαφόρων μέτρων. Επιβεβαιώθηκε λοιπόν στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όντως θα δοθεί επιλογή μεταξύ των αντισταθμιστικών μέτρων προς τον ε, αναφέροντα. Και τέλος, μας ε, ανέφερε ο αναφέροντας ότι όντως έλαβε την επιλογή αυτή. Αυτά λοιπόν όλα μας οδηγούν να θεωρήσουμε ότι η Μάλτα τηρεί την 2005, την 36 του 2005 και άρα επί του παρόντος δεν υπάρχει πλέον ε, παραβίαση της οδηγίας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θετικές εξελίξεις. Θα θέλαμε τώρα να περάσουμε στις αναφορές που έχουν σχέση με τις μεταφορές. Δεν έχουμε αναφερομένους παρόντες, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε αρκετά γρήγορα. Θα δώσω το λόγο στους εκπροσώπους της Επιτροπής. Η πρώτη αφορά ένα κάτοικο της Μάλτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ερώτηση ε, σχετική με την εφαρμογή της προηγούμενης οδηγίας του 1992 για τους περιοριστές ταχύτητας στα λεωφορεία και τα φορτηγά. Η οδηγία του 2002 ε, διευρύνει την υποχρέωση αυτή και στα μικρά λεωφορεία τα οποία έχουν άνω των 9 θέσεων και κάτω των 5 τόνων συνολικού βάρους και στα φορτηγά μεσαίου μεγέθους από 7 μέχρι 12 τόνους γιατί μέχρι τώρα η οδηγία δεν κάλυπτε παρά τα μεγαλύτερα φορτηγά. 1η Ιανουαρίου του 2005 έπρεπε να μεταφερθεί στην Εθνική Νομοθεσία η οδηγία. Η Μάλτα ενσωμάτωσε στην Εθνική της Νομοθεσία την κοινοτική οδηγία τον Οκτώβριο του 2005, ο νόμος δηλαδή του 3, υπαρίθμου 308. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής η μεταφορά θεωρείται πλήρης η Μάλτα χρησιμοποίησε την δυνατότητα εξαίρεσης ε, για τρία χρόνια, μέχρι δηλαδή την 1η Ιανουαρίου του 2008, σχετικά με τα οχήματα τα οποία κυκλοφορούν αυστηρά στο εθνικό της έδαφος. Η οδηγία του 2002 πράγματι προβλέπει ότι οι περιοριστές ταχύτητας τοποθετούνται στα οχήματα από πιστοποιημένες εγκαταστάσεις, πιστοποιημένες από τις εθνικές αρχές. Από πλευράς Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν η μεταφορά είναι πλήρη και δεν υπάρχει καμία διαδικασία επί βάρο βάρος Μάλτα. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη αναφορά είναι ελληνική. Η κυρία Βάγνερ θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ αφορά τον κανονισμό 3577 του 92 του Συμβουλίου σχετικά με τις θαλάσσιες εσωτερικές μεταφορές, το καμποτάζ. Ξεκίνησε μια προσφυγή επί παραβάση εναντίον της Ελλάδος για τη μη προσαρμογή της νομοθεσίας της στις, με, στις μεταφορές ανάμεσα στα νησιά, σύμφωνα με την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης διακίνησης στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών. Υπήρξε μια αιτιολογημένη έκθεση, μια συμπληρωματική για διαδικαστικούς λόγους, στάλει στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι κάποιες πλευρές του καθεστώτος στο οποίο υπέβαλαν τις εταιρείε στον τομέα του εσωτερικού καμποτάζ ήταν αδικαιολόγητες σε σχέση με τους παράγοντες τους οποίους κατά τα άλλα μπορεί να επιβάλλουν με θεμικό τρόπο οι αρχές της χώρας. Μετά από τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπήρξαν σημαντικά βήματα προόδου και έχει, έχει πλέον ε, γίνει συμβατό το εθνικό δίκαιο με το κοινοτικό. Οι γραμμές οι οποίες θα πρέπει να καλύπτονται δημοσιεύονται σε αιτήσια βάση ο έλεγχος του τιμήματος των εισιτηρίων γίνεται με διαφορετικό τρόπο πλέον από τις ελληνικές αρχές οι οποίες φιλελευθεροποίησαν τις γραμμές στις οποίες υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός. Στις γραμμές στις οποίες δεν υπάρχει ένας τέτοιος ανταγωνισμός η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχεται και πάντα είχε αποδεχθεί να υπάρξουν υποχρεώσεις δημόσιων, δημόσιας υπηρεσίας σε σχέση με τον καθορισμό των τιμών. Σε επίπεδο πληρωμάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολύ λιγότερο περιθώρια δράσης. Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του κανονισμού 3577 του 92, για τα σκάφη τα οποία ασκούν καμποτάζ με τις νήσους στο εσωτερικό μιας χώρας, το χώρα είναι θέμα απόλυτα της χώρα υποδοχής, της χώρας δηλαδή στι οποίε διεξάγεται το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Σχετικά με την εσωτερική οργάνωση των σκαφών, οι ελληνικές αρχές προετοιμάζουν ένα νέο προεδρικό διάταγμα, το οποίο έχει σαν στόχο να χαλαρώσει το σημερινό ισχύον του 1999, το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι περιορίζει ιδιαίτερα την ελευθερία κίνησης των εταιριών. Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκονται πάντα σε συζήτηση με τις ελληνικές αρχές σχετικά με τις νομοθετικές υποχρεώσεις που επιβάλλουν στις επιχειρήσεις να κρατούν το δρομολόγιο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, ακόμα και αν υπάρχει κάλυψη στις λεγόμενες άγονες γραμμές, Αναζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρξει μια λύση λοιπόν η οποία να σέβεται τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό αλλά να λαμβάνει υπόψη ε, την ελάχιστη, κατελάχιστον κάλυψη των αναγκών συγκοινωνίας ε, των κοινοτήτων και των κατοίκων που εξακολουθούν να ζουν στα μικρά νησιά. Σας ευχαριστώ πολύ. θα ήθελα να συζητήσω να μην κλείσετε το, μικρό, το μικρόφωνο σας γιατί τα επόμενα πέντε θέματα που έχουν σχέση με τη φορολογία δεν είναι παρόντες οι αναφερόμενοι, εσείς είστε υπεύθυνοι και γι' αυτό δεν ξέρω αν θα πρέπει να σας δώσουμε το λόγο για να δώσετε απάντηση και για τις πέντε. Να μιλήσω αγγλικά σε ό,τι αφορά τις ε, την αναφορά για τον ε, φόρο αναχώρηση στη Μάλτα. Για την πλευρά του φόρου αναχώρηση τώρα. Καταργήθηκε αυτή η επιβάρυνση για τους επιβάτες και από την 1η Νοεμβρίου του 2008 που ξεκίνησε και η χειμερινή σεζόν της ε, αεροπορικής ε. και έτσι στις 27 Νοεμβρίου έκλεισε η υπόθεση αυτή. Εφόσον ο φόρος καταργήθηκε, όλες οι σχετικές καταγγελίες θεωρούμε ότι μπορούν να ε, θεωρηθούν ότι ολοκληρώθηκαν. Σε ό,τι αφορά την τις ε, ναυτικές μεταφορές δεν έχουμε λάβει σχόλια. Θεωρούμε ότι όλα όσα χρησιμοποιήθηκαν για το φόρο αναχώρηση στις αεροπορικές μεταφορές ισχύουν και για τις ναυτικές ε, θαλάσσιες μεταφορές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να εξετάσει το θέμα αυτό περαιτέρω. Ε, σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Κύριε Λό, να αναφέρω ότι επειδή έκλεισε στις 27 Νοεμβρίου του 2008 η διαδικασία επί παραβάση, θα ήταν καλό αν μας είχατε ενημερώσει. Δεν μας ε, ικανοποιεί το γεγονός ότι το μαθαίνουμε μόλις τώρα ένα χρόνο αργότερα ουσιαστικά. Αν θα μπορούσε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας στηρεί ενήμερους σε περίπτωση που ξεκινούν ή κλείνουν περιπτώσεις και διαδικασίες επί παραβάση. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λό ε, για την επισήμανση αυτή, διότι στην Επιτροπή Αναφορών ε, ε, παραπονιόμαστε ότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά, ότι χρειάζεται πολύ χρόνος για να απαντούμε στου αναφερομένους και αν επιπλέον στη μερίσια διάταξη συζητάμε για θέματα που έχουν κλείσει, ε, δεν έχει νόημα. Καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργάζεται έτσι αγαστά μαζί μας. Ευχαριστώ. Κυρία Γκρουνή. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι με αυτό. Σε ό,τι αφορά τις ανοιχτές αναφορές, έχουμε μια ε, γερμανική αναφορά για τις ε, εικαζόμενες παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, απουσιάζει ε, όμως ε, ο αναφερόμενος. Ε, για αναφερόμενη θα ήθελα να ζητήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί. Ε, Κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσω για την αναφορά αυτή, την οποία και υπέβαλε η κυρία Μούλερ. Η κυρία Μούλερ διέμενε στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια. Παντρεύτηκε με Έλληνα πολίτη και αποφάσισαν από κοινού να αγοράσουν ένα διαμέρισμα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, πρώτοι αγοραστές ε, στην Ελλάδα εξαιρούνται από τον πάγιο φόρο της τάξης του 11% επί της αγοράς ιδιοκτησίας. Αλλά στην περίπτωση της αναφέρουσας εξετάστηκε η φοροαπαλλαγή αυτή και δυστυχώς ε, για την αναφέρουσα οι ελληνικές αρχές ζήτησαν ε, να πληρείται άλλος ένας όρος, πέρα από την άδεια παραμονής, να εργάζεται δηλαδή η αναφέρουσα επί ένα έτος τουλάχιστον στην Ελλάδα προκειμένου να δικαιούται την φοροαπαλλαγή αυτή. Ήταν σε άδεια μητρότητας. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι δεν πληρωταν ο όρος αυτός και άρα τη συζήτησαν να καταβάλει το φόρο μεταβίβασης. Ήρθαμε σε επαφή με την αναφέρουσα και ζητήσαμε να μας χορηγηθεί ο σχετικός νόμος βάση του οποίου έδρασαν οι ελληνικές αρχές, τον οποίο και λάβαμε. του 80. Εξετάσαμε λεπτομερός ε, το νόμο αυτό και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο όρος αυτός που θέτουν οι ελληνικές αρχές δεν προκύπτει από τον νόμο. Αλλά δυστυχώς η αναφέρουσα δεν μπόρεσε να παράσχει παρκή αποδεκτικά στοιχεία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να μπορέσουμε να κινήσουμε τη δικασία επί παραβάση και το πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση, δεν δικαιούται καν να εμπλακεί σε διοικητικά ή δικαστικά ζητήματα σε εθνικό επίπεδο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κινήσουμε τη δικασία επί παραβάση, η όρη για την οποία δεν πληρούνταν για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα ενημερώσαμε σχετικά την αναφέρουσα τον Δεκέμβριο του 2008. Μια τελευταία παρατήρηση. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο νόμος αυτός υπόκειται σε μια άλλη διαδικασία επί παραβάση 2007-43-19 και την τελευταία φορά που μιλήσαμε με την Επιτροπή Αναφορών αναφέραμε ότι η διαδικασία, ότι η επιπαραβάση αυτή βρίσκεται σε φάση αιτιολογημένης γνώμης. Οι ελληνικές αρχές δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτά που τους ζητήθηκε και γι' αυτό λοιπόν προσήχθηκε η υπόθεση στο ΔΕΚ το 2009 είναι η υπόθεση C155 του 2009. Και τα στοιχεία τα οποία θεώρησε προβληματικά η Κομισιόν ήταν τα εξής. Καταρχάς, για την εξαίρεση από την, για τη φοροαπολαγή ε, χρειάζεται άδεια μόνιμης κατοικίας, αλλά η Επιτροπή ζήτησε να γίνει διεύρυνση της άδεια αυτής για να συμπεριληφθούν και άτομα τα οποία ζουν στο εξωτερικό και αγοράζουν ε, ακίνητα στην Ελλάδα με σκοπό να εγκατασταθούν εκεί. Γιατί μόνο έτσι τηρούνται οι όροι της ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο στοιχείο, ότι υπό συγκεκριμένου όρους οι Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό και δεν έχουν μόνιμη, άδεια μόνιμης κατοικίας στην ε, Ελλάδα δικαιούνται τέτοια φοροαπαλλαγή, αλλά η φοροαπαλλαγή αυτή σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται σε αλλοδαπούς που δεν μένουν στην Ελλάδα. Και αυτή η διάκριση παραβιάζει την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Για την ενημέρωση αυτή που μας καθησυχάζει. Αυτό σημαίνει δηλαδή τώρα ότι... Α, ο κύριος Γιάρης έτσι το λόγο. Εγώ ε, τα διάκουσα αυτά, αλλά διάβασα και το κείμενο και σκόνταψα σε μία πρόταση που λέει εκεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι πρόκειται για πάγια τακτική της διοίκησης, πράγμα που είναι προϋπόθεση για να ξεκινήσει η προσφυγή επί παραβάση. Και θεωρείται, ας πούμε, μεμονωμένο περιστατικό και δεν μπορεί με βάση ένα μεμονωμένο περιστατικό να ξεκινήσει προσφυγή κατά της Ελλάδας. Δηλαδή ευτυχώς που είχε την τύχη η αναφερόμενη εντό εισαγωγικών να τρέχει μια άλλη παράλληλη περίπτωση στο δικαστήριο και ρωτώ έτσι αφελώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αν αποφασίσει ε, σε μία περίπτωση με μονομένη λάθος η διοίκηση, τι τον νοιάζει τον ενδιαφερόμενο αν είναι πάγια πρακτική, αν του έχει πέσει το κεφάλι μόνο. Το θέμα είναι, είναι ομαδική πρακτική, αν είσαι ένας και σε αφορά εσένα και ένας να είσαι, Αδικήσε. Άρα χάσατε, είναι η απάντηση. Ε, σας λέω ότι είναι αφελής η ερώτηση, δεν ξέρω. Απάντηση. Να τα πω στα γερμανικά, τουλάχιστον να προσπαθήσω. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τα δικαιώματα δηλαδή ενός μεμονωμένου πολίτη να παραβιαστούν από τη διοίκηση, τότε δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ένομα μέσα στη διάθεσή της ε, να παρέμβει, διότι η μοναδική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι βασισμένη στο άρθρο 226 της συνθήκης για τις διαδικασίες προσφυγής επί παραβιάση της ε, συνθήκης. Εμείς δεν μπορούμε να μειχθούμε σε τέτοια πράγματα. Μία εξαίρεση λεγόμενα πιλωτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 15 κράτη-μέλη συμμετέχουν σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, όπου όταν έχουμε μια καταγγελία, όπως αυτή την περίπτωση, τους παραπέμπουμε στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους για να επιληφθεί του θέματος και να απαντήσει στον ενδιαφερομένο εντός 10 εβδομάδων ε, για το πώς ερμηνεύουν την κατάσταση, τι προτίθεται να κάνουν, τι συνέχεια θέλουν να δώσουν για να διορθώσουν αυτή την ε, παραβίαση και να επανορθώσουν. Ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση το πρόβλημα ήταν ότι η Ελλάδα δεν συμμετέχει ακόμα σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Και αυτή λοιπόν η εναλλακτική λύση δεν ε, είναι στη διάθεσή μας προς το παρόν. Ευχαριστώ. Λέει ο Πρόεδρος. Μάλιστα. Ερχόμαστε τώρα στο σημείο Β. Όπως βλέπετε, αναφορές για τις οποίες προτείνεται να περατωθούν υπό το φως της γραπτής απάντησης της Επιτροπής, οπότε δεν χρειάζεται να τις συζητήσουμε και δεν έχουμε τίποτα να πούμε σχετικά. Ένα μόνο θέμα ε, έχω να σας ε, θέσω, να σας ρωτήσω κάτι μάλλον. Ε, έχετε καμία αφιβολία για τη συγκεκριμένη αναφορά, ε, για τις ε, συγκεκριμένες αναφορές. Υπάρχει καμιά αναφορά που θέλετε να ξανανοίξει, αλλιώς θα θεωρήσουμε ότι έχουν κλείσει. Χωρίς μικρόφωνο, κυρία Γιώτοβα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για την αναφορά υπαριθμών 41. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό για μας, που είναι η μοίρα ε, κάποιων παιδιών με πνευματική αναπηρία, ε, ορφανών, εγκαταλελειμμένων στη Βουλγαρία. Πέρυσι, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του Κοινοβουλίου, ε, υπήρξε ένα ντοκιμαντέρ ε, του καναλιού BBC4 για ένα τέτοιο ίδρυμα ορφανοτροφείου στη Βουλγαρία. Δεν το λέω επειδή είμαι Βουλγάρα, αλλά επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ ε, καιρό, πάρα πολλά χρόνια με το θέμα αυτό, ε, θέλω να το θέσω προ συζήτηση. Η απάντηση που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μεν ικανοποιητική, αλλά εγώ επιμένω να μην κλείσει αυτή η αναφορά για να μπορέσουμε ε, του χρόνου να κάνουμε επιτόπου, μάλλον να ζητήσουμε επιθεώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτόπου σε συνεργασία με τις βουλγαρικές αρχές για να δούμε κατά πόσο έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα ή λύνεται στη Βουλγαρία. Δυστυχώς το θέμα αυτό έχει ε, γίνει πλέον μεγάλη ε, ιστορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγιναν εκδηλώσεις και εδώ στο Κοινοβούλιο σχετικά. Και αν ενδιαφέρεται κανείς, ε, ακόμα μπορούμε να σας δώσουμε για επιπλέον εξηγήσεις και υλικό. Παρακαλώ όμως να μην κλείσει προς το παρόν, να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και να ε, μείνει υπό παρακολούθηση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Νομίζω ότι όλοι μας είδαμε το ντοκιμαντέρ αυτό, το οποίο μας ε, σόκαρε όχι μόνο σε ό,τι αφορά την Βουλγαρία, αλλά και άλλες χώρες. Τώρα, για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε, να ζητήσω τη γνώμη της Γραμματείας. Κάθε μέλος, λέει η Γραμματεία, έχει δικαίωμα να ζητήσει να παραμείνει ανοιχτή μία αναφορά. Εφόσον λοιπόν το ζητήσατε, θα παραμείνει ανοιχτή. Να σας πω ότι υπάρχουν πολλές αναφορές για το θέμα αυτό και στην τελευταία θητεία έγινε και μία διερευνητική αποστολή επιτόπου. Επισκεφτήκαν ε, ένα από τα ιδρύματα αυτά και άρα υπάρχει και μία σχετική έκθεση η οποία διατίθεται στα μέλη της Επιτροπής και αναφέρει πιο πολλές λεπτομέρειες για το θέμα που ε, μας παρουσίασε η κυρία Ρόντεβα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Αυτή τη διαδικασία θα ακολουθήσουμε λοιπόν. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ολοκληρώσαμε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πέρα τη συνεδρίασης και σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας.